Colleagues, Λοιπόν, παρακαλώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε πάπυρον. Έχουμε και την προσκεκλημένη μας. Όσοι δεν πήγαν σήμερα στην Κοπενχάγη, περιμένουν να έρθουν, ελπίζω να έρθουν. Γιατί θα έχουμε μία συζήτηση σε ό,τι αφορά τη με εξωτερική μελέτη για τα εμπόδια πρόσβασης των υποψηφίων στα διαρθρωτικά ταμεία. Πολύ σημαντική μελέτη που έρχεται και σε πολύ επίκαιρο χρονικό σημείο αφού συζητούμε και το πολιτές πλαίσιο. Θέλουμε να περιορίσουμε τους φραγμούς στη χρηματοδότηση για τα επόμενα χρόνια και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα ζητήσω λοιπόν από την κυρία Χάμζα να κάνει την παρουσίαση καταρχάς και ελπίζω στη συνέχεια να έχουμε και μια ανταλλαγή απόψε. Να ευχαριστήσω και το Φρανς που της κρατάει παρέα της κυρίας Χάμσα. Α, άλλη έβλεπα, με συγχωρείτε, είστε εσείς που είστε δίπλα μου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα σας μιλήσω για τα εμπόδια των υποψηφίων σε τεφά την πρόσβασή τους στα διαρθρωτικά ταμεία. Μου είπαν ότι είναι λίγο μακροσκελή παρουσίαση, οπότε είτε θα παρακάψω κάποιε διαφάνειε, είτε θα τι διατρέξω γρήγορα. Καταρχάς να σας δώσω το υπόβαθρο αυτής της μελέτης. Δεν υπάρχει μια συνεκτική εικόνα, είναι προφανές αυτό, ε, της ε, πρόσβασης στα διευθυντικά ταμεία, α, αυτών. Και ούτε και η κοινή γνώμη γνωρίζει πολύ καλά ε, τα σχετικά. Πριν ξεκινήσω με τα πορίσματα και τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, θα ήθελα να σας ε, εξηγήσω διορισμούς. Πρώτον όρος beneficiaries, δικαιούχοι και applicants υποψήφοι. Κάποιες φορές ε, στα κείμενα προκύπτουν δυσκολίες ανάλογα και με το είδος της χρηματοδότησης σχετικά με το TST δικαιούς και το TST ετών. Δικαιούχος είναι ουσιαστικά το πρόσωπο το οποίο παίρνει τη χρηματοδότηση και ο ετών είναι αυτός που κάνει την αίτηση για τη χρηματοδότηση ήδη ε, δικαιούχων. Δημόσιες αρχές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, φυσικά πρόσωπα, ιδίως ε, στο ESF, το Κοινωνικό Ταμείο και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα γιατί στο Τζέρεμι και το Τζέσικα δικαιούχοι είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τελικούς δικαιούχους τις εταιρείε, την εταιρεία, την εκάστοτε η οποία ε, αναλαμβάνει την ε, υλοποίηση ενός έργου την μελέτη μας την έχουμε βασίσει στον κύκλο διαχείρισης προγραμμάτων, διότι πιστεύουμε ότι σε καθένα από τα τέσσερα στάδια αυτού του κύκλου υπάρχουν ζητήματα τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν, να, να αποτελέσουν εμπόδια τέλο πάντων για τους υποψηφίους. Ας ξεκινήσουμε τη φάση του προγραμματισμού πρέπει να είναι μια διαδικασία απλούστερη και πιο εύκολη για την πρόσβαση των υποψηφίων. Μετά έχουμε και την ε, υλοποίηση, την ε, παραγωγή, τη δημιουργία του σχεδίου και τέλος τη διαχείριση. Αυτά είναι τα τέσσερα στάδια. Τέσσερα επίπεδα έχουμε διακρίνει. Εκεί βλέπουμε κάποιους ε, παράγοντες που επηρεάζουν. Πρώτο επίπεδο το ευρωπαϊκό. Εδώ έχουμε τις αρχές τερικής σχέσης, τους κανονισμούς και ό,τι διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα περίοδο. Δεύτερο επίπεδο για μας το σημαντικότερο σε σχέση με τους υποψηφίους φυσικά το εθνικό επίπεδο, διότι τα διαθροτικά ταμεία, τα μέσα της πολιτικής συνοχής εδράζονται, βρίσκονται στο εθνικό και τοπικό επίπεδο και πραγματικά πολλές φορές εκεί ανακύπτουν πραγματικά εμπόδια. Τρίτο επίπεδο, επίπεδο προγράμματος όπου τα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικό τρόπο το ένα από το άλλο. Αυτό βέβαια πάντοτε εξαρτάται από το σχεδιασμό, αλλά μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο ή όχι τον υποψήφιο. Και τέταρτο επίπεδο, το επιχειρησιακό, όπου οι διαδικασίες των υποψηφίων, διάδοση κτλ. τα ε, περιλαμβάνονται σε αυτό το επίπεδο και υπάρχει και ένα τελευταίο επίπεδο, το επίπεδο του έργου, του project του ίδιου που έχει να κάνει με την πλέον, με την ικανότητα του ε, δικαιούχου ή του ετούντος σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Στο εθνικό επίπεδο οι σημαντικότεροι παράγοντες είναι προφανώς η συγχρηματοδότηση που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό ιδίως εν καιρό κρίσης και δεύτερον τα διοικητικά συστήματα Ανάλογα με τα διοικητικά συστήματα που έχουν τα κράτη-μέλη, αν είναι δηλαδή ομοσπονδιακά, αν έχουν αναργανωμένα κεντρικά, ανάλογα με αυτά λοιπόν τα συστήματα λειτουργεί και διαφορετικά και το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Οι άλλοι δύο είδη τύποι παραγόντων που επηρεάζουν είναι η δυνατότητα διαχείρισης προγράμματος, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, διότι βλέπουμε να υπάρχουν πολλά προβλήματα στα κράτη-μέλη στον τομέα αυτό, ε, λόγω διακυμάνσεων στο προσωπικό. Και το σύστημα δημοσιονομικής στήριξης, οικονομικής στήριξης μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Και τρίτοι παράγοντες, επιχειρησιακοί παράγοντες, δηλαδή διάδοση των πληροφοριών, διαδικασία της υποβολής αίτηση, επιλογής ε, και μετά την ανάθεση διαχείριση. Σε πολλές περιπτώσεις οι αιτούντες δεν υποβάλλουν εκ νέου αίτηση γιατί θεωρούν ότι η διαδικασία μετά την ανάθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη για αυτούς. Γι' αυτό βάζουμε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό. Τώρα, παράγοντες οι οποίοι απαντούν στα διάφορα επίπεδα, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στρατηγικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο και προϋπολογισμός των διαφορετικών ταμείων. Οι κανονισμοί στην προκειμένη περίπτωση τροποποιήθηκαν στη διάρκεια της περίοδου προγραμματισμού περιλαμβάνουν την αρχή της εταιρική σχέσης, απαιτήσει ενημέρωση πληροφόρηση, την οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση και τι απλουστεύσει που σα είπα. Παράγονται σε εθνικό επίπεδο, όπω ήδη προείπα, το θεσμικό διοικητικό σύστημα έχει μεγάλη σημασία για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Επίσης, η διάθεση των πόρων που μπορεί να είναι είτε παράλληλη προς τα εθνικά προγράμματα είτε να είναι ενοποιημένοι, γιατί αυτό κάνει και μια διαφορά. Και επίσης έχουμε και την ρευστότητα, την εθνική και την περιφερειακή για τη συγχρηματοδότηση. Παράγονται σε επίπεδο διαχείρισης. Εδώ έχουμε τη δομή και τις ικανότητες, δυνατότητες, με βάση την ιεραρχική δομή, δηλαδή ανάλογα με το πόσα ιεραρχικά επίπεδα υπάρχουν. Εάν αυτοί που διαχειρίζονται το πρόγραμμα έχουν τις ικανότητες προς αυτό. Κάποιες φορές δεν ισχύει, δεν είναι ικανή. Και έπειτα έχουμε το σύστημα οικονομικής υποστήριξης. Κάποιες επιδοτήσεις ε, που δεν επιστρέφονται ή κάποια δάνεια που πρέπει να επιστραφούν κτλ. Παράγονται σε επιχειρησιακό επίπεδο, σε αυτό επικεντρωνόμαστε κατά βάση. Έχουμε την επιλογή των διαδικασιών υποβολής αίτησης, πληροφόρηση, διάδοση, στήριξη των δικαιούχων, είδη, συστήματων ε, ε, ε, έτσι και τα λοιπά. Στα πράσινα βέλη που βλέπετε τώρα εδώ, αναφέρονται ε, στα ζητήματα που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα και στις συνετεύξεις που πραγματοποιήσαμε, διότι δεν υπάρχει και πολλή βιβλιογραφία για αυτά τα θέματα. Επομένως, κάναμε συνεντεύξεις σε 90 επιχειρησιακά προγράμματα ανά την Ευρώπη ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των συνεντεύξεων. Πρώτα απ' όλα, τα είδη των διάβλων ενημέρωση. Τα βλέπουμε σε όλο τον κύκλο. Ξεκινά πολύ απλά από τα διαφημιστικά σποτ, από τα τηλεοπτικά σποτ, ε, κάποια περιοδικά, στην φάση του προγραμματισμού, ιδίως στα κράτη-μήλου που υπάρχει μεγάλος προϋπολογισμός για το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ένα παράδειγμα είναι η Πολωνία, όταν έχει μεγάλη σημασία για, την, για το συγκεκριμένο παράδειγμα χάρη πρόγραμμα. Ε, όταν έχουμε την υλοποίηση, ε, οι ιστοσελίδες είναι πολύ σημαντικό. Κάποιες φορές δεν τις ε, επικαιροποιούν, ε, δεν είναι προσαρμοσμένες στις ε, εξελίξει των πρώτη των εργασιών και όταν ο ετών βλέπει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των, δια, των επικοινωνιακών αυτών διάβλων, αποθαρρύνεται και δεν ε, αναζητά την χρηματοδότηση. Ε, και επίσης η εθνική χρηματοδότηση σε αρκετές ε, δυτικοευρωπαϊκές χώρες είναι και ευκολότερη και λιγότερο πολύπλοκη. Και αν αυτό ισχύει και υπάρχουν και περισσότερες πληροφορίες τότε θα είναι και πιο εύκολη και η υλοποίηση του σχεδίου. Μετά στην παραγωγή του σχεδίου, στην δημιουργία του, στην εκτέλεσή του, ε, τα email, τα σεμινάρια, κάποιες εκδηλώσεις δηλαδή ενημερωτικέ είναι σημαντική διάβλη παροχής πληροφοριών και στη φάση της διαχείρισης του προγράμματος οι διμερείς επαφές και συνομιλίες. Σχετικές πτυχές λοιπόν ε, στους διάβλους επικοινωνίας και ενημέρωσης. Το είδος του μέσου ποικίλει ανάλογα με το πρόγραμμα. Στα προγράμματα υποδομών δεν χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν συγκεκριμένοι διάβλοι γιατί λίγοι είναι μόνο οι αιτούντες. Παραδείγματο χάρη στην Αυστρία έχουμε τρεις εργολάβους ε, για εργαδοποίηση, οπότε δεν χρειάζεται να ε, δοθούν ε, πληροφορίε σε ένα ευρύ φάσμα ετούντων. Υπάρχουν προγράμματα όμως που χρειάζονται διαφορετικούς διάβλους επικοινωνίας σε περισσότερες της μιας γλώσσες και πιο εξατομικευμένα. Όταν υπάρχει ευρύ φάσμα ε, ετούντων υπάρχουν και πολύ και διαφορετικοί διάβλοι. Ποια είναι τα δύο βασικά εμπόδια με τους διάβλους παρέχεις πληροφοριών. Αυτά δήλωσαν οι ετούντες τουλάχιστον. Είναι η έλλειψη εναρμόνισης, ιδίως στις ιστοσελίδες. Είδαμε στην περίπτωση της Ιταλίας συγκεκριμένα ότι η ιστοσελίδα του επιχειρησιακού προγράμματος έχει διαφορετικές πληροφορίες από την κρατική ιστοσελίδα. Δεύτερον, έλλειψη κατάλληλων πληροφοριών. Ε, οι δυνητικοί ετούντες ή ετούντες δεν βρίσκουν καν πού πρέπει να απευθυνθούν για να ε, υποβάλουν την αίτησή τους. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι των συνεντεύξεων είχε να κάνει με την ε, διαδικασία της υποβολής αίτησης. τα οικονομικά ζητήματα, για να το πω απλά, είναι το σημαντικότερο ζήτημα. Και δεύτερο, το διοικητικό άχθος. Τρίτον, είναι οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί, που δυστυχώς δημιουργούν πιο πολλά προβλήματα από αυτά που αρχικά φανταζόμασταν ότι θα δημιουργούσαν. Χρηματοοικονομικά ζητήματα. Έλλειψη κατάλληλης ε, εθνικής χρηματοδότησης. Αυτό ισχύει κυρίως για όσα κράτη-μέλη δεν έχουμε αναλογία της ε, ευρωπαϊκής με την εθνική χρηματοδότηση σε χώρες με μικρό περιπολογισμό διαρθρωτικό. Όταν δεν γίνονται πολλές προσπάθειες για την προσαρμογή, την αντιστοίχηση των δύο ειδών χρηματοδότησης. Δεύτερο πρόβλημα, έλλειψη προ-χρηματοδότησης. Ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, είναι χρονοβόρα διαδικασία η υποβολή της και οι μικρές επιχειρήσεις πολλές φορές έχουν πρόβλημα να βρουν πόρους και να ε, χρηματοδοτήσουν ε, την διαδικασία υποβολής αίτησης. Και η χρήση εξωτερικών συμβούλων επίσης είναι ένα ζήτημα. Και γι' αυτό απαιτούνται χρήματα, όπως και για την προηγούμενη διαδικασία της υποβολής της αίτησης. Στο ρυθμιστικό πλαίσιο πρώτα απ' όλα βλέπουμε δυσκολίες ε, σε ό,τι αφορά τους κανόνες της κρατικής ενίσχυσης. Ουσιαστικά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα εδώ όσο είναι με τους εθνικούς κανόνες ε, των δημοσίων προμηθειών. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δηλαδή απαιτεί ε, από τους υποψηφίους αρχικά να σέβονται τους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες. Και όταν προσπαθεί μετά ο διαχειριστής του έργου να εκτελέσει το έργο θα πρέπει να εφαρμόσει κανόνες κρατικών προμηθειών. Εκεί βλέπουμε να υπάρχει πρόβλημα για τους project managers, τους διευθυντές των έργων. Επίσης, άλλο πρόβλημα, ότι αλλάζουν συχνά οι κανόνες να αλλάζει δηλαδή ο κανόνας ε, μέσα στην ε, φάση της εκτέλεσης του έργου. Και έτσι ο διευθυντής του έργου ασχολείται με αυτές τις αλλαγές και δεν ενημερώνται σωστά υποψήφοι ετούντες. Τρίτο θέμα, διοίκηση, διαχείριση και υποστήριξη. Πολυπλοκότητα ήταν μια λέξη που την ε, ακούσαμε σε πάρα πολλές συνεντεύξεις. Όπως και την ε, φράση έλλειψη σαφών κατευθυντηρίων γραμμών, έλλειψη σαφών κατευθύνσεων. Δηλαδή, οι εκτελεστικοί φορείς δεν έχουν ε, σαφή καθοδήγηση και τελικά δεν ξέρουν στην πράξη τι πρέπει να κάνουν. Τα έγγραφα τώρα που πρέπει να παρασχεθούν πολλές φορές είναι και αυτά πολύπλοκα και κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να παράσχουν όλες αυτές ε, τις ε, δηλώσεις, όλα αυτά τα έγγραφα. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι ο διαθέσιμος χρόνος. Οι υποψήφοι, οι ετούντες μάλλον, παραπονούνται θεωρώντας ότι το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή αιτήσεων, ο ένας μήνας δηλαδή, είναι σύντομος και δεν επαρκεί για να υποβληθεί μια πλήρης αίτηση. Επίσης δεν είναι παρκή τα επίπεδα διαφάνειας και συνεκτικότητας. Αυτό τι θα πει ότι δεν είναι πολύ κατανοητό το γιατί πήρε ένας υποψήφιος, ένας ετών ε, κάποιο κονδύλι και ένας άλλος όχι. Δεν είναι καθόλου σαφές. Έλλειψη σαφήνειας σχετικά με την επιλεξιμότητα και ο διευθυντής του έργου ε, και οι εκτελεστικοί φορείς δίνουν ε, πληροφορίες στους ετούντες, δίνουν όμως αντιφατικές πληροφορίες και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει επίσης επαρκή στήριξη από τους εκτελεστικούς φορείς και επίσης επειδή υπάρχει ανακύκλωση προσωπικού συχνά, ε, δεν υπάρχει επαρκής τεχνογνωσία και επαρκής ικανότητες. ιδίω στα νέα κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν κίνητρα για το προσωπικό για να παραμείνει στη θέση του για μακροχρονικό διάστημα, δεν είναι ε, πολύ καλή μισθή και έχουμε συχνά αυτά τα φαινόμενα ανακύκλωσης, ε, μετακίνησης του προσωπικού. Οπότε χάνεται και η σχετική τεχνογνωσία. Για τα προγράμματα ETC υπάρχουν άλλα θέματα διαφορετικής φύσεως. Πρώτα απ' όλα, αναζήτηση εταίρων Εκεί χρειάζονται τουλάχιστον ένα ή δύο εταίροι, τουλάχιστον, και δεν υπάρχει πολλές φορές επιθυμία διασυνοριακής συνεργασίας. Το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ο γλωσσικός φραγμός. Άλλα, άλλα θέματα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η απουσία εμπιστοσύνη μεταξύ δημοσίων αρχών, κρατικών αρχών και ετούντων. Διαπιστώνουμε ότι πιστεύουν ότι δεν θα έχουν εμπιστοσύνη στον project manager οι δημόσιες αρχές. Επίσης δεν υπάρχει η νοοτροπία η επιχειρηματική της κίνησης δηλαδή μιας νέας επιχείρησης. Φερρυπίν, άκουσα ότι ιδιαίτερα οι μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, δεν έχουν τέτοια νοοτροπία και Βέβαια, εν τέλει, η οικονομική κρίση είναι ένας από τους κύριους λόγους που αντοπίζονται αυτή την εποχή. Ορισμένα Είναι ένας τρόπος λοιπόν που έχουν ε, να αντιμετωπίσουν οι αρχές ε, είναι με πρακτικές που προλαμβάνουν τα προβλήματα προσπαθούν να προχρηματοδοτήσουν οι δυνατόν. Σε ορισμένε περιπτώσει όμω αναγκάστηκαν και λόγω εθνικών ή άλλου, ε, άλλης προελεύσεως διατάξεων να σταματήσουν αυτή την προχρηματοδότηση. Ε, ή αλλιώς υπάρχουν ζητήματα σε σχέση με τις τράπεζες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν έχοντας καλή γνώση και γνώση του χώρου και έτσι μπορούμε να προσφύγουμε σε αυτές. Μια άλλη λύση που είχαμε δει Φερρυπίν στην Αυστρία ήταν το One Stop Shop, όπου δηλαδή τα εθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα έδειξαν την καλύτερη αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των προγραμμάτων και λεπίδραση μεταξύ των διαφορών ε, ε, χρηματοδοτικών μέσων. Η τελική φάση είναι αυτή στην οποία θα πρέπει ο ετών να καλύψει τη δαπάνη. Μόνο στο βέβαια που πρέπει να αποφεύγεται γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό ή διαφορετικά θα πρέπει να επέμβει ε, μια επαγγελματική οργάνωση όπως ένα εμπορικό επιμελητήριο για να στηρίξει οικονομικά τον ετούντα ε, πράγμα το οποίο συμβαίνει σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι μετά την ε, έγκριση υπάρχουν πάλι προβλήματα. Έχω, α πούμε, περίπτωση ενό ετούντο ο οποίο είπε ότι μετά την έγκριση διαπίστωσε ότι είναι τόσο πολλέ δυσκολίε που δεν πρόκειται να ξαναυποβάλει τέτοιε προτάσει. Προβλήματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με την φάση μετά την ε, έγκριση. Καθυστερήσει τις πληρωμές. Όπως είπα, ήδη πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία του ε, σχεδίου χωρίς την πληρωμή, η οποία μπορεί να λάβει χώρα και ένα χρόνο αργότερα, πράγμα το οποίο είναι αφόρητο βάρος οικονομικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, είναι πολύ συχνά ε, ιδιαίτερα περίπλοκος και χρονοβόρος ο τρόπος, οι διαδικασίες γενικότερα διοικητικές που προβλέπονται και η απόδοση των οικονομικών λογαριασμών. Το έχουν επισημάνει πολύ αυτό. Τρίτον, απουσία εμπιστοσύνη, το να με αυτό νωρίτερα. Επίσης αισθάνονται μερικές φορές ότι αντί να τους υποστηρίζουν οι αρχές που ελέγχουν, μάλλον, τους, ε, μάλλον έχουν αστυνομική δράση. Πράγμα το οποίο είναι λάθος ασφαλώς. Θα πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα να ε, τη χάνουν εμπιστοσύνης οι κανόνες σχετικοί με τις δημόσιες προμήθειες επίσης, που έχει εγκρίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελούν ένα άλλο πρόβλημα. Η απουσία ευελιξίας ως προς τον επαναπροσδιορισμό επαναδιαπραγμάτευση στόχων. Δεν μπόρεσαν δηλαδή να ξαναπροσαρμόσουν στις ανάγκες ένα σχέδιο μετά την έγκριση του. Αντιλαμβάνονται κατά τα άλλα όμως τις παρατηρήσεις τους ε, οι αιτούντες ότι είναι απαραίτητη παρακολούθηση και η επαλήθευση ότι τηρούνται οι όροι. Επίσης τώρα, σε σχέση με την απλούστευση και τις τροποποίησεις. Δεν έχουν ε, υλοποιηθεί, δεν έχουν ε, μάλλον γίνει δεκτές με θετικό τρόπο όλες οι προσπάθειες απλοποίησης ή απλούστευσης. Δεν δηλώνουν όλοι δηλαδή υπέρ της απλούστευσης, γιατί η Φερρυπίν έγινε κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περίοδου η απλούστευση και έτσι ο διαχειριστής του προγράμματος, ο project manager, δεν ήθελε να ξαναρχίσει να ε, ε, αναπροσαρμόζεται σε, νέες, σε νέους κανόνες. Επίσης, project manager ή program manager μπορεί να έχει δώσει θετική κρίση για την ε, απλούστευση, αλλά ταυτόχρονα επισημένοντας ότι το κατά το ελάχιστο ποσοστό του 20% είναι πολύ χαμηλό και έτσι δεν, αρκεί. Αν και πρέπει να επισημάνουμε ότι οι περισσότεροι από τους ετούντες δεν είχαν επαρκείς γνώσεις για τις προσπάθειες απλούστευσης ή διαπίστωναν ότι δεν τους έλυναν προβλήματα, δεν αφαιρμόζονταν δηλαδή σε εκείνους αποτελεσματικά γιατί είχαν να κάνουν με χρηματοδότηση ε, περισσότερο υπερσυνοριακών προγραμμάτων εξωτερικών συνόρων, ειδικότερα Φερρυπίν σχέσεις με βαλκανικά κράτη υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και το μεγαλύτερο ποσό του ενδιαφέροντος των εθνών. Και έτσι δεν είχαν ε, εφαρμογή στις περιπτώσεις αυτές οι επιλογές επιλοποίησης. Συμπεράσματα. Η διάθεση της συγχρηματοδότησης είναι ο πιο σημαντικός ε, παράγων, διαθεσιμότητα της συγχρηματοδότησης. Το λένε οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες, ε, ωστόσο ότι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτος ο τρόπος με τον οποίο αναγνωρίζεται η δυνατότητα αυτή, και τη δυνατότητα αυτή. Επίσης, απουσία ικανότητας υλοποίησης ε, απουσία δυναμικού στα, στις, ε, στους φορείς υλοποίησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, άρα χρειάζεται αυτή να ενισχυθεί. Τα διαρθρωτικά ταμεία πάλι που είναι σωματωμένα στα εθνικά συστήματα χρηματοδότησης. Τα εθνικά δηλαδή και τα ευρωπαϊκά συστήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν καλύτερα, να ευθυγραμμιστούν καλύτερα το ένα στο άλλο. Αυτό τουλάχιστον στην Αυστρία έχει ήδη προχωρήσει. Και δυσκολίες που εμφανίζονται μόνο όταν ε, στοχοποιείται ένα μικρό ποσοστό ή ένας μικρός περιορισμένος αριθμός δικαιούχων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη, οι πληροφορίες που προσφέρονται είναι πολύ πιο περιορισμένες. Άλλα συμπεράσματα, ε, σχέδια, έργα που έχουν να κάνουν με το εισόδημα παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες διότι δεν έχουν την ικανότητα να ε, χειριστούν τέτοια σχέδια, τέτοια έργα δηλαδή, οι αρμόδιες αρχές ή επίσης ο δικαιούχος ο οποίος ε, έχει να κάνει με μέτρα καινοτομίας πολλές φορές αντιμετωπίζει δυσκολίες για λόγους προστασίας ευρεσιτεχνιών και ούτω καθεξής και έτσι πολλοί είναι αυτοί οι, μικρο, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν θέλουν να ζητήσουν τη χρηματοδότηση προκειμένου να αποφύγουν την υποχρέωση για δημοσίευση της εφεύρεσής τους ή της καινοτομίας τους. Το ίδιο σε σημαντικό βαθμό αντιμετωπίζουν και τα πανεπιστήμια και οι ιδιωτικοί φορείς ε, στις εταιρικές, σε εταιρικέ σχέσεις με πανεπιστήμια και ιδιωτικούς φόρους. Επίσης προβλήματα έχουμε ως προς τις ιδιαίτερες προκλήσεις ή τους γλωσσικούς φραγμούς. Συστάσεις μας εν ολίγης. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να χορηγηθούν ε, ευέλικτα ποσοστά χρηματοδότηση, δηλαδή τα ποσοστά που διατίθεται αυτή τη στιγμή προβλέπονται από την νομοθεσία πρέπει να αναθεωρηθούν. Επίση θα πρέπει να ενισχυθεί η υλοποίηση των ε, μέσων δημοσιονομικής μηχανικής με περισσότερη ευελιξία. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια μέσα μένα, αλλά πολλοί είναι οι project manager οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύ περίπλοκα και έτσι τα αποφεύγουν. Τρίτον, θα πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση, η εφαρμογή της χρηματοδότησης για τις μικρούς, ε, μικρής κλίμακας δικαιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Θα πρέπει να περιοριστούν οι κίνδυνοι τέταρτον από δημοσιονομικές διορθώσεις. Οι διορθώσεις δηλαδή της δημοσιονομικής διαχείρισης στο τέλος του project δεν έχουν νόημα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι εκφράζουν την, ε, το, στόχο, το στόχο ή το τέλος του ε, έργου. Επομένως θα πρέπει να τροποποιηθούν. Και πέμπτον θα πρέπει να ενισχυθεί η σε πρώιμο στάδιο αποζημίωση. Δηλαδή, όπως επεσήμανα νωρίτερα, έχουν πρόβλημα ως προς την χρηματοδότηση του πρώτου, πρώτου έτους του έργου οι δικαιούχοι. Έκτον, θα πρέπει να διατηρηθεί η γενική λογική και η δομή των διαστροτικών ταμείων. Υπάρχουν ε, πολλοί ε, δικαιούχοι και υποκράτη κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ε, ως προς την προσαρμογή στους νέους κανόνες και τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν κατά καιρού. και έτσι θα πρέπει η γενικότερη λογική, η ορολογία ή κάποιοι γενικοί όροι να διατηρούνται απαράλλακτοι ε, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να καταλαβαίνει όταν αλλάζει κάτι τι έχει αλλάξει και να παρακολουθεί τους κανόνες. Επίσης, όποιες αλλαγές θα πρέπει να εισάγονται στην πρωταρχική φάση του προγράμματος. Πολλές φορές έχουν εισαχθεί στα μισά του προγράμματος και έτσι δεν έχουν εφαρμοστεί σε ορισμένα κράτη-μέλη. Επίσης, τυποποιημένα έγγραφα, που είναι ένα ακόμα ζήτημα που επισημαίνουν ε, και αυτό το βλέπουμε διότι δεν μπορεί να υπάρχει συγκρισιμότητα μεταξύ των εκθέσεων περί υλοποίησης Ιδιαίτερα δε οι δαπάνες του κώδικα της Λισαβόνα μεταξύ κρατών μελών δεν είναι συγκρίσιμες. Συνεχίζω με τις συστάσεις. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αποτελέσματα, σε μια διαδικασία που θα οδηγήσει αποτελέσματα, τερολογική δηλαδή. Θα πρέπει να ενισχυθεί η ανταλλαγή πείρας και γνώσης. Διαπιστώνουμε επί παραδείγματι ότι δεν αποστέλλονται σε πολλές περιπτώσεις οι project manager από τα κράτη-μέλη σε ε, σεμινάρια ανταλλαγής εμπειρίας διότι ε, λαμβάνεται υπόψη το κόστος αυτής της αποστολής. Επίσης θα πρέπει ενδεχομένω να αναθεωρηθεί ο ορισμός των μικρομεσαίας επιχείρησης. Υπάρχουν επιχειρήσεις με 250 εργαζομένους οι οποίες ε, χάνουν την το χαρακτηρισμό της ε, δικαιούχου μικρομεσαίας επιχείρησης, αλλά δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε και ως μεγάλες επιχειρήσεις, στους φερρυπίν τράπεζες και το καθεξής και έτσι, δεν μπορούν ούτε σε αυτές να συγκαταλευθούν και να ωφεληθούν από χρηματοδότηση ε, ούτε στα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βέβαια. Επίσης θα πρέπει ε, προγραμματικά μέτρα για την καινοτομία να επαναπροσδιοριστούν, να επανεξεταστούν, διότι όπως είπα ε, διστάζουν οι ενδιαφερόμενοι να δείξουν καινοτομία ή να ε, αποκαλύψουν στοιχεία της καινοτομίας τους, της τους, ε, του δημιουργικού τους πνεύματος σε τέτοια προγράμματα. Και γι' αυτό δεν μπαίνουν στα προγράμματα. Άλλη σύσταση, καλύτερη εμπλοκή των εταίρων στη στρατηγική ανάπτυξη διότι βλέπουμε ότι μερικές φορές ε, η παρουσία εταίρων είναι απλώς ένα άλοθη, είναι ένα προπέτασμα και στην πραγματικότητα αποφασίζει ο Υπουργός ακόμη σε πολλές περιπτώσεις άνωθεν τι θα ε, γίνει. Βελτίωση επίσης πέραν των ε, ειδικών συνθήκων ή που μπορεί να ισχύουν σε μια χώρα, βελτίωση των συστημάτων ενημέρωσης, πληροφόρησης, να μην υπάρχουν δύο-τρεις διαφορετικές ιστοσελίδες για το ίδιο θέμα. Ε, ένα σύστημα ευέλικτο και διαφανές για την λειτουργία, για τον έλεγχο, για την παρακολούθηση, γιατί όπως είπα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι αισθάνονται ότι ε, τους παρακολουθούν ε, αστυνομικές αρχές ε, η επανεξέταση των δημοσίων των κρατικών προμηθειών είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει βέβαια να απασχολήσει τα κρατημέλη. Τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν ε, με το ευρωπαϊκό όριο, γιατί μερικά κράτη-μέλη έχουν ε, κανονισμούς που αναφέρονται σε 500 ευρώ το πολύ. για κάθε αγορά. Ε, επομένως, είναι περί, περιπλοκή πιστεύω αυτός ε, τέτοιου είδους κανόνες και βέβαια εμποδίζει την αξιοποίηση, την απορρόφηση δημόσιας χρηματοδότησης. Επίσης ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μπορεί να ξεκινάει σε ένα Υπουργείο και να ξεκινάει κανεί εκεί να κάνει την εκπαίδευσή του και μετά να έρχεται μια ιδιωτική επιχείρηση για να πάρει το ίδιο αυτό προσωπικό το οποίο έχει καταρτιστεί με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να το προσλάβει με τριπλάσια αμοιβή. Αυτό δεν θα πρέπει βέβαια να γίνεται. Επίση, κάτι το οποίο διαπιστώνουμε σε κράτη-μέλη με μεγάλο ε, προπολογισμό. Για τα μία ταμεία λόγιστα μικρότερα είναι αυτό. Και συστάσεις για το εθνικό περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αποστέλλονται ή προσφέρονται μηνύματα ενημέρωση, πληροφόρηση συνεπιστο στην προκατακτική όσο και στην ύστερη φάση. Δηλαδή πριν να ξεκινήσει κανείς ένα σχέδιο έχει λάβει μία πληροφόρηση και στη συνέχεια να αντιλαμβάνεται ότι δεν ισχύει πια τίποτα ή ασχύουν διαφορετικά πράγματα. Επίσης η έννοια της μονοθυριδικής προσέγγισης, στο λεγόμενο one-stop shop που έχουμε ήδη στην Αυστρία, αλλά που είναι απαραίτητο να υπάρξει παντού, δηλαδή να υπάρχει ένας, ένας χώρος στον οποίο θα μπορεί κανείς να απευθυνθεί και επίσης θα μπορεί μέσω αυτού του χώρου να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο ίδιο πρόγραμμα. Η διάχυση ε, παραδειγμάτων καλής πρακτικής, βέλτιστης πρακτικής. Θα μπορούσαμε δηλαδή να ενισχύσουμε την ε, κοινοποίηση των ενδιαφερόμενων, στον ετούντα, ε, παραδειγμάτων βέλτισης πρακτικής, ώστε να διευκολύνουμε τη δουλειά του. Ε, η απλούστευση των διαδικασιών για υποβολή αίτησης πρέπει να αναπτυχθεί σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό συγγνώμη και περιφερειακό επίπεδο. Μέχρι στιγμής γίνεται σε εθνικό επίπεδο, δεν εφαρμόζεται όμως όλα τα προγράμματα. Η... Ε, αρχές που έχουν σχετική εμπειρία πρέπει προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία της προετοιμασίας αυτών των αιτήσεων να συμμετάσχουν πιο ένεργα. Ακόμα δεν γίνεται αυτό. Καλύτερη ο σχεδιασμός της διαδικασίας των προτάσεων, της υποβολής των προτάσεων. Στην αρχή, Φερρυπίν, ένας μήνας που μερικές φορές προβλέπεται στα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι δεν αρκεί για την προετοιμασία μιας πρότασης. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας αφιερώσετε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάμσα. Φαντάζομαι ότι μπορούμε να πάρουμε και την παρουσίασή σας για να την ε, διαβιβάσουμε και σε όλους τους συναδέλφους. Θέλω τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους για την υποβολή ερωτήσεων ή σχολείων. Η μελέτη σας πραγματικά είναι συναρπαστική. Λαμπέρ, βλέπω ότι είσαστε έτοιμος ήδη να πάρετε το λόγο να αρχίσετε πυροβολείτε. <laughs> Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κοιτάξτε, είναι μια κρίσιμη χρονική στιγμή αυτή, αυτή την εβδομάδα. Ε, οι συνάδελφοι μπορούν να κάνουν τα τελευταία σχόλια που θα ληφθούν υπόψη για τραπέζι το του κανονισμού, αν άκουσα καλά. Πολλά ελήφθαν υπόψη ε, στην ε, εκπόνηση του νέου κανονισμού. Οπότε το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον ε, τελικά λείπουν πράγματα. Είναι δύσκολο να τα εντοπίσει κανείς τα κενά, διότι όπως είπατε και εσείς, πολλά πράγματα ελήφθησαν υπόψη. Είναι δύσκολο όμως τελικά ποια είναι τα κενά ποια, έχουν, ε, ποια στοιχεία έχουν υποπέσει τη προσοχή μας. Οπότε επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια. Σε ό,τι αφορά την ε, προχρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτό το έχουμε καταγράψει ως ένα πραγματικά μείζον ζήτημα. Αν είχε σε μη καπαόμικρον και ξεκινάς ένα μεγάλο project, 400.000 ευρώ για παράδειγμα. Εντάξει, δεν είναι τεράστιο το μέγεθο για μα, όμω είναι μεγάλο το ποσό για μια μη κυβερνητική οργάνωση που θέλει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα σε μια τοπική κοινότητα. Οπότε, όταν μιλάμε για προχρηματοδότηση, στο παρελθόν οι περιφερειακέ αρχέ είχαν ένα κάποιο ταμείο από όπου προβλεπόταν η προχρηματοδότηση. Τη σημερινή στιγμή αυτό δεν συμβαίνει πλέον είναι κάτι που πρέπει να καταγράψουμε. Και εξ όσων γνωρίζω και σε κάποιου άλλου τομεί πολιτική, θέλω να πω ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα προχρηματοδότηση. Παρακαλώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αυτό πρέπει να γίνει σωστά. Είναι κάτι σημαντικό δεν έχουμε ενδιαφερόμενους, γιατί δεν έχουν, αν θέλετε, κονδύλια κίνησης, τα 20.000 ευρώ για να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία και δεν, δεν υπάρχει βοήθεια από τις τράπεζες. Ε, Τέλειωσε η εποχή των παχαίων αγελάδων. Τώρα, για τις καθυστερημένες ε, πληρωμές. Κάτι περίεργο σημαίνει εδώ, διότι χθε ακούσαμε ότι σε 10 κράτη-μέλη έχουν μπλοκαριστεί ε, σε μεγάλο βαθμό πολλές πληρωμές. Κάποιοι συνάδελφοι είπαν ότι αυτό οφείλεται ίσως στην έλλειψη ε, ρευστού από την Κομισιόν και άρα εντοπίζει όλο και πιο πολλούς λόγους και αφορμές για να μπλοκάρει χρηματοδότηση. Αυτό είναι καταστροφή. Σε αυτό το πεδίο πολιτικής ε, θα πρέπει να κάνουμε κάτι, να είμαστε πιο αξιόπιστοι, διότι στα πλαίσια μιας νέας συνεργασίας, ίσως στη νέα δημοσιονομική περίοδο, θα δούμε μεγάλη προθυμία από τους ενδιαφερόμενους. Θεωρώ λοιπόν πρακτικός πώς πρέπει να ε, κρατούμε κάποια επίπεδα αξιοπιστίας ε, στην συνεργασία μας και στο πώς καταβάλουμε και εμείς πληρώμες από πλευράς Ένωσης. Είπατε κάτι τώρα άλλο. Αν το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν αλλάξουν, τροποποιούν έναν κανονισμό, οι πρακτικές δεν αλλάζουν αντίστοιχα στις χώρες. Δηλαδή, τι κάνουμε. Κατά τη διάρκεια μία ε, θητεία του Κοινοβούλου μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδου ε, συνεχεί τροποποιήσει. Άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον από εσά. Α πάρουμε το παράδειγμα τη Ρουμανία, για παράδειγμα, για το, τα θέματα στέγαση ε, και τα θέματα οικοδομή για ευάλωτε κοινωνικέ ομάδε ο σχεδιασμός της χρήσης των διαθροτικών ταμείων και της κοινή διαχείρισης είναι κάτι που απαιτεί έναν προγραμματισμό με ορίζοντα ενό ή δύο ετών, γιατί ε, η διεθνωτική πολιτική λειτουργεί σε ορίζοντα χρόνου. Σε μία λοιπόν χρονική στιγμή κρίση, σε μία χρονική στιγμή που επιθυμούμε να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε άμεσε επενδύσει ε, κομμένε και ραμμένε ε, στι ανάγκε, ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τι θέσει εργασία και σε μια πιο πράσινη οικονομία, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αλλάζουμε. Αν αλλάζουμε συνθήκες, αν απαιτείται, να μπορούμε να αλλάζουμε. Όπως κάναμε πριν από κάποιο διάστημα, όταν απευθύναμε μια έκκληση στα κράτη-μέλη να ε, δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην απασχόληση των νέων. Και σήμερα τι ακούμε, χθες από ό,τι ακούσαμε, 5 έως 8 διοχετεύονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα για την απασχόληση των νέων. Οπότε τίθεται το ερώτημα. Πιστεύετε ότι μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα σύστημα ξεκάθαρο σχετικά με τις θεματικές του προτεραιότητες ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να συνάπτονται και συμβάσει εταιρική σχέση, αλλά ταυτόχρονα να κρατούν και επαρκή ευελιξία. Θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει κατά κύριο λόγο να συζητήσουμε είναι να λάβουμε υπόψη τις πραγματικές ανάγκες ε, των επιχειρήσεων, των πανεπιστημίων κτλ. και να προσαρμόσουμε τα εργαλεία μας. Οπότε ρωτώ. Ε, Βάσει μελέτη σα, θεωρείτε ότι μπορούμε μέσα στο πλαίσιο που κινούμεθα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Και τι συγκεκριμένε ιδέε θα μπορούσαμε να καταθέσουμε, πώ νομίζετε εσεί ότι μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Κοιτάξτε, καλό θα ήταν αυτή η μελέτη να έρθει ένα μήνα νωρίτερα. Πάντω θα ψηφίσουμε τον Ιούλιο και πιστεύω ότι στον Ιούλιο θα μπουν πολλά στο τραπέζι από του συναδέλφου. Πιστεύω ότι πραγματικά λάβατε υπόψη πολύ καλά project και αυτή η μελέτη λέει πολλά. Δίνει πολλές προοπτικές ε, στον θέμα της χρηματοδότησης και της κοινή διαχείρισης ε, των περιφερειακών ε, project. Από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως προβλέπεται η χρηματοδότηση δημόσιο του τομέα και άρα μπορούν να γίνουν τέτοιου διευθετήσει σε επίπεδο κρατών μελών. Ίσως τελικά να μακρηγόρησα. Ίσως θα μπορούσατε όμως να μου απαντήσετε και να μου δώσετε μια εικόνα. Ευχαριστώ, ε, Λαμπέρ. Ο κύριος Νίλσον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τρία σχόλια από πλευρά μου. Ζητώ συγγνώμη, δεν ήμουν παρόν να ακούσω όλη την παρουσίαση, γιατί έπρεπε να ψηφίσω μια άλλη επιτροπή. Έλαβα χθε την ε, παρουσίαση, την ε, μελέτη, συγγνώμη, και διάβασα προσεκτικά τα συμπεράσματα. Πρώτο σχόλιο. Συμφωνώ με τον κύριο Λαμπέρ. Πολλά εκ των συστάσεων ήδη έχουν ληφθεί υπόψη από τους συγκητές μας. Αυτό είναι θετικό. Δεύτερον, σε κάποιο σημείο της μελέτης μιλάτε για συστάσεις σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Μιλάτε για ευρωπαϊκή ανταλλαγή. Αυτό είναι σημαντικό και μπορούμε να έχουμε μια τέτοια ανταλλαγή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε, τη δική μου εμπειρία στη Βόρεια Σουηδία, η εμπειρία από project άλλων χωρών ήταν πραγματικά ε, μείζονο σημασία. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να στηρίζουμε τέτοιου είδου ανταλλαγέ εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τρίτο και πιο σημαντικό, πολύ σημαντικό για την απόφαση της Επιτροπής μας, λέτε ότι απευθύνεται σε συστάσεις σε τέτοιο επίπεδο καλύτερη συμμετοχή των εταίρων στη στρατηγική κατάρτιση ε, των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική συμμετοχή, πρακτική συμμετοχή των εταίρων. Αυτή είναι και η δική μου εμπειρία. Ξέρετε, έχω γνωρίσει δύο περιφέρειες σε αυτή την προγραμματική περίοδο στη Σουηδία, όπου η μία περι, περιφέρεια. Εκεί είχαμε τη μαρτυρία ε, έντονη συμμετοχή των εταίρων ευθύ εξ αρχή για την δημιουργία του προγράμματο και η υλοποίηση έγινε πολύ καλύτερη. Στην άλλη περιφέρεια, αντίθετα, ο περιφερειάρχης ουσιαστικά τον έλαβε όλο μόνος του και δεν είχαμε συμμετοχή των εταίρων άρα η... και καταλήξαμε στην υλοποίηση σε πολύ μικρότερο βαθμό. Αν θέλετε λοιπόν επιτυχία, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των εταίρων από την αρχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σίμων. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και διεξοδική η παρουσίαση που μας δείχνει ότι θα πρέπει να διαφοροποιούμε μεταξύ διαφορών σημείων που μπορούμε να επιλύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί όπου μπορούμε δηλαδή να διαμορφώσουμε τα διαφορετικά ταμεία, αλλά και προβλήματα τα οποία είναι εσωτερικής φύσεως, που προκύπτουν στα ε, ε, κράτη, μέλη, και ως εκ τούτου πρέπει να επιληθούν σε αυτά. Ένα πράγμα λοιπόν το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε, για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο, θα ήταν να είναι πιο υποχρεωτική, πιο δεσμευτική συμμετοχή των ε, εταίρων στα προγράμματα όπως εκτελούνται στην κάθε χώρα. Γιατί εάν θέλει κανείς μια συγχρηματοδότηση, αν ζητήσει συγχρηματοδότηση με στόχο την ανάπτυξη ενός σχεδίου, αλλά πάντα με συγχρηματοδότηση, τότε θα πρέπει να δίνει το σχέδιό του, το χρονοδιάγραμμά του κτλ. Αλλά εάν ένας δυνάμει εταίρος ενδιαφέρεται μεν, αλλά δεν μπορεί. Φέρει πριν μια δημοτική αρχή. Δεν μπορεί για διάφορου λόγου ε, να συμμετάσχει, γιατί δεν έχει μέσα στο μεσοπρόθεσμό τη ε, δημοσιονομικό σχεδιασμό προβλέψει τα κονδύλια αυτά με τα οποία θα έπρεπε να συμμετάσχει, τότε θα έπρεπε να υπάρχει ε, κάποια λύση. Νομίζω αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, διότι συνήθως ή συχνά δεν είναι τόσο το πρόβλημα το ποσό της χρηματοδότησης αλλά το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να προβλέψει το ποσό αυτό, να δεσμεύσει το ποσό αυτό. Και εδώ υπάρχουν πολλές φορές διατάξεις κρατικές ενδεχομένω, οι οποίες δεσμεύουν τις ε, αρχές και δεν τους επιτρέπουν να ε, διαθέσουν ε, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τα ποσά αυτά, να τα έχουν προβλέψει ήδη στον προπολογισμό τους. Ευχαριστώ κύριο Χρυσόγελος από ό,τι βλέπω στα ετολόγο και κανείς άλλος, έτσι είναι. Θέλει κανείς άλλος. Ο κύριος Χρυσόγελος, παρακαλώ. Ναι, νομίζω ότι και στη συζήτηση που κάνουμε εδώ για τα διαρθρωτικά ταμεία ε, δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση πράγματι στο ρόλο της αναβάθμισης των ικανοτήτων των ε, φορέων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, οι φορείς οι οποίοι θα κάνουν έτσι ή θα συμμετάσχουν στο σχεδιασμό πρέπει, πρέπει να έχουν αυξημένε ικανότητε για να μπορεί να πράγματι να αξιοποιηθεί το εργαλείο από τα χρηματοδοτικά ταμεία. Ε, θα έλεγα επίση ένα πολύ σοβαρό θέμα από την εμπειρία μου σε περιφερειακό επίπεδο είναι ότι πολλέ φορέ σχεδιάζονται έργα τα οποία κατασκευάζονται, υλοποιούνται, αλλά δεν έχει προβλεφθεί πραγματικά, παρά μόνο τυπικά, η βιώσιμη λειτουργία ή διαχείριση του έργου. Να σα αναφέρω ένα παράδειγμα. Ε, είναι πολύ συχνό στη χώρα μου να φτιάχνεται ένα βιολογικό καθαρισμό, Αλλά μετά δεν έχει προβλεφθεί η μακροχρόνια λειτουργία αυτού του βιολογικού καθαρισμού και με αποτέλεσμα να έχει επενδυθεί κεφάλαιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και ο βιολογικό καθαρισμό να τίθεται εκτό λειτουργία και να μην επιτελεί το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε. Άρα είναι πολύ σημαντικό στα προγράμματα να δοθεί έμφαση στο αποτέλεσμα και στη συνέχεια τη λειτουργία των έργων και μετά την ε, ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. Αυτό θα γλιτώσει και χρήματα από του φορολογούμενου, αλλά και σίγουρα θα ε, δώσει έμφαση σε αυτό που θέλουμε να επιτελούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή πραγματικά οι υποδομές αυτές να λειτουργούν μακροχρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάμσα θα ήθελε να σχολιάσει. Όσα ακούστηκαν. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι υποστηρίζω τα λεγόμενα του Γερμανού ε, βουλευτή. Πράγματι. Ε, είναι θέμα σωστής διαχείρισης και χρήσης των ευρωπαϊκών κανονισμών. Εκείνη η ουσία. Για παράδειγμα, η ενοποίηση των κανονισμών για τις δημόσιες προμήθειες κάτω από τα ευρωπαϊκά κατόφλια θα μπορούσε να είναι μια προσέγγιση. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η συμμετοχή των εταίρων. Ήδη απαιτείται η συμμετοχή τους. Το πρόβλημα είναι ότι τα Υπουργεία το κάνουν πολύ επιφανειακά. Καλούν τους εταίρους σε μια συζήτηση στην αρχή του project, μετά ε, τους καλούν να προσυπογράψουν το project και τελείωσε. Καμία ανταλλαγή ουσιαστικής, αν θέλετε, συνεισφοράς προτάσεων. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι μπορεί να γίνει. Οι κανονισμοί είναι νέοι αν κάποιοι ξεκίνησαν κάποια project την τελευταία προγραμματική περίοδο και έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν αυτά τα εργαλεία, τώρα πρέπει να κάτσει στα θρανία πάλι και να ξαναδιαβάσει. Ε, διότι υπάρχει το θέμα της γεωργίας και της αλίας ε, στα εργαλεία κοινωνικής συνοχής λαμβάνουν πώ λοιπόν τα εργαλεία συνοχή στη γεωργία και την αλληλεία. Οπότε θα πρέπει να ξανακάτσουν οι ενδιαφερόμενοι να διαβάσουν πώ θα έχουν τη συνεργασία, την κατάλληλη συνεργασία ανάμεσα στα εργαλεία. Τώρα, η ανταλλαγή εμπειριών, τα προγράμματα ETC προβλέπουν μια κάποια διάδραση, interaction. Και δεν έχει δώσει κακά αποτελέσματα αυτή η διάδραση. Όσοι λοιπόν ε, συνεργάζονται στα πλαίσια μίας ε, διεθνικής συνεργασίας ε, έχουν μια τακτική επαφή και επικοινωνία. Θα μπορούσε λοιπόν αυτή η πλατφόρμα επικοινωνίας, αυτή η διάδραση, το Interact αν θέλετε, μπορεί να αποτελέσει μοντέλο και για άλλου είδους project. Τώρα, για την ανάπτυξη δυναμικού. Το πρόβλημα εδώ έγκυται στο εξή. Όταν έχουμε μία οικοδόμηση δυναμικού, αύξηση δυναμικότητας, Το θέμα είναι πώς θα χειριστεί αυτή τη δυναμικότητα και πού θα δώσει μετά ε, το βάρος αυτούς που του έχει δοθεί μεγαλύτερη δυναμικότητα και πού θα στοχεύσει. Εντάξει, υπάρχουν πολλά που βοηθούν. Ε, ένας καλύτερος μισθός είναι ένα δέλεαρ. Μιλάμε για χώρες όπου άνθρωποι που εντάσσονται σε αυτά τα project δεν παίρνουν πάνω από 300 ευρώ το μήνα, οπότε δεν είναι ένα δέλερ για να ε, καθίσει κανείς μακροπρόθεσμα και να αφοσιωθεί στη ζητήματα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, αγαπητοί συναδελφοί, θα κλείσω αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή εδώ. Αν κατάλαβα καλά θα μας δώσετε την παρουσία σας, γιατί πραγματικά ε, είχε δώσει, έχει δώσει πολύ καλά στοιχεία, καθώ επισημάνεται τα πλέον ακαθόδη ζητήματα στο όλο θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας και να πω στους συναδέλφους ότι αν έχετε και άλλες ερωτήσεις, μπορείτε μέσω της γραμματείας να έρθετε σε επαφή ε, με την κυρία Χάμσα και με τους ε, συνεργάτες που εκπώνησαν αυτή τη μελέτη. Σας ευχαριστώ. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μποστινάρου. Ταμείο Συνοχής και κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου 1084-2006. Βίκτορ, θα σου δώσω το λόγο και μετά θα δώσω το λόγο στους ε, σκιώδεις και στους λοιπούς συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Μισή ώρα έχουμε στη θέση μας για αυτή την έκθεση. Ελπίζω να μην ξεπεράσουμε το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ αρχής να σας πω ότι θα είμαι απολύτως προβλέψιμος. Η γνωμοδότησή μου για την έκθεση και η προσέγγισή μου είναι γνωστές. Τώρα θα ήθελα απλώς να παρουσιάσω κάποια νέα στοιχεία που διαπιστώνω στο τελευταίο χρονικό διάστημα, που έχω συμπληρώσει δηλαδή και βεβαίως περιμένω να ακούσω πάνω από όλα τα σχόλιά σας. Καταρχάς, οι νέες τροπολογίες έχουν να κάνουν περισσότερο με την ε, διασύνδεση των Δημοτικών Ταμείων με το Euro Facility. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να περιμένουμε, να διαγράψουμε τα ποσά και να περιμένουμε να γίνει διαπραγμάτευση η σχετική με τα ποσά και τότε να τα συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας. Δεν υπάρχει λόγος να συζητούμε για ποσά όταν ακόμα δεν είναι αυτά ε, ε ξεκάθαρα. Για να είμαστε και σε συνέπεια με την έκθεση για το Γενικό Κανονισμό και ελπίζω να σας αρέσει η πρότασή μου. Επίσης, Και εδώ μιλάμε για τα 10 δις, έτσι, που θα γίνει μεταφορά. Για τα κριτήρια που θα ισχύουν για τα ποσά που ίσως να μεταφερθούν, σημειώνω ότι τα ποσά αυτά μπορούν να εφαρμοστούν αποκλειστικά και μόνο σε έργα του Ταμείου Συνοχής στα κράτη-μέλη, και το Ταμείο Συνοχή, τα δαπάνε του πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Συνοχή. Επίση, μιλούμε για κριτήρια που θα πρέπει να υλοποιεί μια, να εφαρμόζει μια κεντρική υπηρεσία ή κεντρική υπηρεσία κατά την επιλογή των ε, επιλέξιμων προγραμμάτων ή έργων. με ιδιαίτερη έμφαση στο να αποφεύγεται η αδίποτε στρέβλωση στις αρχικές εθνικές προτάσεις στον εθνικό φάκελο. Άρα αυτό που λέω ότι κατά τα τρία πρώτα χρόνια της προγραμματικής περίοδου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2016 η επιλογή των έργων θα γίνεται με πλήρη σεβασμό των εθνικών ε, ποσών, των ποσών που αντιστοιχούν στο κάθε κράτο μέλο, που έχουν μεταφερθεί από το Ερωτικά στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχή και έτσι. Κάθε κράτη, τα κράτη-μέλη θα έχουν επαρκή χρόνο για να προετοιμαστούν, για να σχεδιάσουν, για να προτείνουν ε, έργα και να αναπτύξουν ε, την θεσμική και διοικητική δομή που χρειάζεται. Μετά την 1η όμως Ιανουαρίου του 2017 θα είναι πλήρως λειτουργικό με τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό ε, αυτών, το European Facility. και επίσης προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη συνοχή ε, με το Διευθυντικό Ταμείο στο βαθμό που αφορά περισσότερο θέρμανση ε, και παραγωγή ενέργειας. οι δε μονάδες, οι λεγόμενες, ε, οι, οποίες μπορούν να ξεπεράσουν τα 20 ΜΒ, το λεγόμενο powerhouse δηλαδή, θα πρέπει να ε, ελέγχεται ότι είναι συμβατές έτσι ώστε και να αποκατασταθεί η λειτουργία τους, να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση λειτουργίας και να μην ξεπερνούμε τις ε, ε, προβλέψεις των έργων. Μόνο λοιπόν πάνω από 20 ΜΒ θα χρηματοδοτούνται και όπου χρειάζεται θα γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής θερμότητας και τουρμπίνων, τουρμπινών με το σχετικό δίκτυο διανομής. Το Ταμείο Συνοχής δηλαδή θα ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και θα παρακολουθεί με τους χρονικούς περιορισμούς ολόκληρο τον κύκλο της παραγωγής θερμότητας, της διανομής και της χρήσης της ενέργειας μέσα σε κτίρια αναμορφωμένα. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών και σχετικών πηγών ενέργειας δεν θα έχουν προβλήματα χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Για δε τις λοιπές τροπολογίες που κατατέθηκαν ήδη στο πρώτο ε, σκαρίφημα δεν θα ήθελα να ε, γρηγορήσω, να χρονοτριβήσω περισσότερο, αλλά θα υπογραμμίσω μόνο το εξή. Ότι η αποτελεσματικότητα χρήση ενέργεια στην στέγη, στην οικιακή στέγη, είναι για το Ταμείο συνοχή ένα από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους και οικονομικούς τρόπους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας χρήσης ενέργειας και της επίτευξης των στόχων της, ε, του, του 2020. Γνωρίζουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από άλλους ε, φορείς, από άλλες πηγές, ότι έχει μεγάλη βραδιπορία σημειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους στόχους του 2020 και αν υλοποιηθούν αυτά τα οποία προτείνω εγώ, πάλι μόνο 10% θα έχουμε επιτύχει. Άρα θα έχουμε, σημαντική, ε, θα έχουμε σημειώσει μια σημαντική ήταν θα έλεγα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, δεν έχουμε μόνο τους στόχους του 2020. Θέλουμε να ενισχύσουμε την πράσινη διάσταση της οικονομίας μας. Θέλουμε να βελτιώσουμε το ενεργειακό μείγμα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες μα επιχειρήσεις. Θέλουμε ριζικά να περικόψουμε τις ε, εκπομπές του του άνθρακα. Και θέλουμε να καταστήσουμε την ενέργεια που θα πληρώνει ο πολίτης πιο οικονομική για την τσέπη του. Και πρέπει να σας πω ότι στο Βουκουρέστι, την πρωτεύουσα της πατρίδας μου, συναντήθηκα με εμπειρογνώμονες, με επιστήμονες ε, που ασχολούνται ιδιαίτερα με την, ε, ηλεκτρική, με την ηλιακή ενέργεια. Αν λοιπόν στο σύστημα και με τις γεωθερμικές πηγές, Αν λοιπόν στο σύστημα της θερμότητας ενταχθούν και η γεωθερμική και η ηλιακή πηγή ενέργειας, τότε όχι δεν βελτιώνεται, αλλά μειώνεται η απόδοση της ενέργειας κατά 40%. Χωρίς δηλαδή την αποκατάσταση, την αναμόρφωση Χωρί την εξοικονόμηση ενέργειας. Κατά 40% πράγμα το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ υψηλό. Θα έχουμε λοιπόν 40% εξοικονόμηση και μόνο από αυτό. Ταυτόχρονα έχουμε και την αποτελεσματικότητα στην χρήση ενέργεια και το 36% από περικοπή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επιπλέον η αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργεια πρέπει να προωθηθεί από το Ταμείο Συνοχής, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει επιπλέον σημαντικό ρόλο για ορισμένε περιφέρειες λόγω των διαφόρων ε, κριτηρίων επιλεξιμότητας σε σχέση με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και πρέπει το Ταμείο Συνοχής βέβαια να ανοίξει και για άτομα με αναπηρίες και για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος της ε, ε, διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, τη Σύμβαση των Ηνωμένων και άρα πρέπει να προσαρμοστούμε στι διεθνεί μα υποχρέωσει. Η αρχή επίση ο πληρώνει πρέπει να ενσωματωθεί πλήρω στο Ταμείο συνοχή και στη λειτουργία του. Ε, πάντως σημαντικό είναι το μήνυμα αυτό, όπως να θέλω να ανοίξω τη συζήτηση, να διευρύνω υπερβολικά τη συζήτηση, πρέπει να απευθυνθεί το μήνυμα αυτό στον Επίτροπο Ποτόπνικ, Πρέπει να βρει δηλαδή ο ίδιος τρόπο να διατυπώσει εκ νέου το κείμενο της προτάσεις, ώστε αυτή η αρχή ορυπαίνων πληρώνει να εφαρμόζεται πλήρως και από το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Συνοχής να είναι ανοιχτό σε πρόσβαση μόνο σε μια ε, κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άκρος έκτακτης ανάγκης και όχι σε καθημερινή βάση, για να μην ανατρέπεται η αρχή ο πληρώνει. Για δε το Natura 2000 θα ήθελα να ενισχύσω την πτυχή της προστασίας της βιοποικιλότητας μας, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της δυνατότητας για επιλεξιμότητα έργων που σχετίζονται με το Natura 2000. Η συμπερίληψη του περιβάλλοντος της Natura μαζί με εκείνο του Urban μπορεί με τρόπο συνεπή, συνεκτικό με τρόπο ολιστικό να καλύψει τους δύο τομείς του urban και μαζί με, το urban, ε, με τους χώρους του urban 1 που τους ή άλλως έχει μεγάλη σημασία για την, ε, είναι ένα θεμελιώδες ε, έργο και ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινή μας ζωή. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει και η κινητικότητα του κοινού να είναι ε, ένας από τους στόχους, ε, παράλληλα με το Urban 1, για να μειωθεί και η περιβαλλοντική ρήπανση και η ε, μεγάλη κίνηση στους δρόμους, η συμφόρηση, η κυκλοφοριακή και ούτω καθεξής. Επίσης θέλω να ευχαριστώ τον συνάδελφο που κατέθεσε μια τροπολογία όπου ζητούσε για τους κοινούς δείκτες, οι κοινοί δείκτες των έργων να ε, προχωρούν μέσα από τις εκτελεστικές πράξεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι από την νομοθεσία της θα υπάρχει περισσότερη ευελιξία και η προσαρμοστικότητα σε νέε συνθήκε, οι οποίε φανταζόμαστε θα διαφέρουν πολύ από τώρα σε μερικά χρόνια. Μετά το 2014 μπορούμε να έχουμε νέε διαστάσει να προβλέψουμε νέες ζεστάσεις εμείς Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ επίσης όλους τους συναδέλφους τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής ε, για τη συνεργασία, όλους τους συναδέλφους και για τις ε, για τη συμβολή τους στο έργο και βεβαίως θα προσπαθήσω να ενσωματώσω στη τελική έκθεση κάθε προσφορά κάθε πρόταση και τροπολογία συναδέλφων. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι αύριο στις 6 το απόγευμα. Παρακαλώ λοιπόν, μην ξεχάσετε να καταθέσετε τις τροπολογίες σας και σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Μόνο ο Νίκος Χρυσόγελος είναι εδώ σκιώδης, έχετε το λόγο. Ε, I would like to thank Mr. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουστινάρου. Ας μιλήσω ελληνικά. I'd like to thank you, Mr. because... Uh, Θέλω να σας ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου, είχαμε πολύ επικοδομητική συνεργασία. Και θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας ε, για να βελτιώσουμε την ήδη καλή πάντως έκθεσή σας, που πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Yes, ε, μερικές τροποποιήσεις, μερικές προσθήκες. Νομίζω ότι η έκθεση Μποστινάρου είναι σε καλή κατεύθυνση, σε σωστή κατεύθυνση. Οι, οι προτάσεις μας είναι κυρίως στην κατεύθυνση να, γίνει, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ του χρηματοδοτικού εργαλείου και των ε, απαιτήσεων για ε, αηφορία και να είναι συνεκτική η χρηματοδοτική πολιτική με τους στόχους της Ευρώπης 2020, της στρατηγική 2020. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα στο θέμα των έργων ε, που έχουν σχέση με τις μεταφορές, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σήμερα το 90% όλων των μετακινήσεων με ιδιωτικά γεωταχή αφορά αποστάσεις μέχρι 6 χιλιόμετρα. Και αυτό βέβαια συνεισφέρει στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ε, ε, αερίων του θερμοκηπίου. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε έμφαση σε εκείνες υποδομές που είναι πιο βιώσιμες, που είναι πιο συμβατές με τους στόχους μας για την μείωση των κλιματικών ε, επιπτώσεων και της ε, προστασίας του κλίματος. Θέλουμε λοιπόν όλα τα έργα να ε, μειώσουν τις εξωτερικές, το εξωτερικό κόστος, το external cost. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πάμε ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με αυτό που ξέραμε ως χρηματοδοτήσεις μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι απλώς να φτιάξουμε υποδομές, αλλά να κάνουμε εκείνες υποδομές, εκείνα τα έργα που οδηγούν προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Και γι' αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για νερό, για απόβλητα ή για ε, έργα μεταφορικά, πρέπει να επιλέξουμε τις προτεραιότητες μας. Και αφού έχουμε πολιτικές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα νερά, για, τις, ε, για τα απόβλητα, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε εκείνα τα έργα που ανταποκρίνονται στην ιεραρχία. Για παράδειγμα, μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για επαναχρησιμοποίηση, μιλάμε για ανακύκλωση όχι μόνο των απορριμμάτων, αλλά μιλάμε και για τα θέματα του νερού. Μέχρι τώρα η έμφαση, για παράδειγμα, είναι στο τέλο τη διαδικασία να επεξεργαζόμαστε τα λίμματα. Αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση νερού ε, μέσα στα δίκτυα, μέσα στι κατοικίε, μέσα στου επαγγελματικού χώρου. Άρα πρέπει να ανεβάσουμε ε, τι προτεραιότητε αυτέ και στα θέματα της χρηματοδότησης. Επίσης, πολύ σωστά και στην έκθεση αναφέρονται ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα, καθώς και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα θέματα επίσης των μεταφορών πρέπει να τονίζουμε συνεχώς ότι μιλάμε για βιώσιμες μεταφορές και όχι απλώς για μεταφορές. Άρα μετατοπίζουμε το ενδιαφέρον και τις χρηματοδοτήσεις προς τα συστήματα που είναι πιο βιώσιμα. Επίσης θα, ε, πρέπει να πούμε ότι ε, εμείς τουλάχιστον ως πράσινοι είμαστε υπέρ του να μειωθούν τα έργα ε, κατασκευής μεγάλων οδικών αξώνων εκτός αν συμβάλλουν στις διασυνοριακές συνδέσεις. Όπως επίσης δεν μπορεί να χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους αεροδρόμια τα οποία βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 200 χιλιόμετρα από άλλο υπάρχουν ε, αεροδρόμιο. Δηλαδή πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τις υποδομές συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για, ε, για, για κατοικίες, κυρίως, όχι κυρίως μόνο στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ε, εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λένε στο μέσος μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τον Ίσκε και τον εισηγητή, έχει πολύ σημαντικά ωφέλη, όχι μόνο περιβαλλοντικά και ενεργειακά, αλλά και οικονομικά. Σε μια εποχή κρίσης, είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν οι λογαριασμοί, ειδικά για τα νοικοκυριά, τα οποία αποφέρουν πολύ από χαμηλούς μισθούς ή από την ανεργία. Άρα λοιπόν είναι ένα κατάλληλο εργαλείο να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση, όχι μόνο σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο ε, ενέργειας και περιβάλλοντος. Ε, Επίσης πρέπει να δώσουμε στα θέματα της προστασίας του κλίματος και της προσαρμογής κλιματικές αλλαγές μεγάλη έμφαση σε υποδομές που αναβαθμίζουν το ρόλο των οικοσυστημάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πολλές μελέτες, πολλές έρευνες που δείχνουν ότι μπορούμε και το κλίμα να το προστατεύσουμε και να, να δημιουργήσουμε τείχους άμυνας απέναντι στις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές, βελτιώντας το ρόλο, αναβαθμίζοντας το ρόλο των οικοσυστημάτων. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, άρα εδώ πρέπει να το τονίσουμε στην έκθεση ιδιαίτερα ε, και να το κάνουμε και πράξη μέσα από τις ε, χρηματοδοτήσεις. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό, όπως έχει τονιστεί σε όλη τη συζήτηση που κάνουμε εδώ στην Επιτροπή, ότι ο ρόλος των διαφόρων κοινωνικών φορέων, της αυτοδιοίκησης, τοπικής και περιφερειακής, της κοινωνίας των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός. Αυτός ο ρόλος για να είναι αποτελεσματικός πρέπει να βασίζεται σε καλή γνώση και στην προετοιμασία και στο σχεδιασμό και στην παρακολούθηση υλοποίηση και στην αξιολόγηση. Άρα πρέπει να, πράγματι να δώσουμε έμφαση στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων αυτών των φορέων, ε, ειδικά για τη δικιά μας χώρα, την Ελλάδα, και σαν πράσινη έχουμε καταθέσει μια πρόταση, ειδικά αυτή τη στιγμή που η κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ε, αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτός ο ρόλος να περάσει πολύ άμεσα, να βρούμε έναν τρόπο να περάσει άμεσα στις περιφέρειες και στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε πράγματι τα χρήματα που υπάρχουν και το λέμε συνέχεια, τα 14 δις και παραπάνω χρήματα ευρωπαϊκά που υπάρχουν για να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη τη Ελλάδα και να δημιουργηθούν θέσει εργασία, να περάσει μέσα από τι περιφέρειες και του Δήμου. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό και για το μέλλον, όχι μόνο χωρών σαν την Ελλάδα, αλλά και άλλων χωρών, ειδικά των νέων κρατών μελών. Δηλαδή να ενδυναμώσουμε την ικανότητα, τη γνώση και την δυνατότητα να παίξουν σημαντικό ρόλο οι περιφέρειες και η αυτοδιοίκηση, ουσιαστικά οι τοπικέ κοινωνίε, τα έργα, είτε άμεσα είτε και έμεσα, Όταν σχεδιάζεται ένα έργο για την περιοχή του να έχουν λόγο, καθοριστικό, όχι απλώ τυπικό, το ακούσαμε και πριν, αλλά και να μπορούν να είναι σε θέση να ε, υλοποιούν, να αξιολογούν, να αλλάζουν, να τροποποιούν και να σχεδιάζουν. νομίζω αυτά είναι. Ε, είμαστε έτοιμοι, έχουμε καταθέσει σε γενικές γραμμές τις παρατηρήσεις και τελειώνω μόνο λέγοντας ότι και στους δείκτες πρέπει να βελτιώσουμε τους δείκτες που περιγράφουν αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Δεν αρκούν, όπως λέγαμε, απλώς χιλιόμετρα δρόμων ή κυβικά μέτρα ε, νερού, πρέπει να περιγράφουμε ακριβώς και την διαφοροποίηση που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε παράδειγμα να συγκεντρώνουμε το νερό της βροχής, πρέπει να έχουμε ένα δείχτη που να λέει τι ποσοστό είναι αυτό στη συνολική κατανάλωση νερού. Αν θέλουμε να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση του νερού μετά το βιολογικό καθαρισμό, πρέπει να έχουμε δείκτες που να ξέρουμε ότι πράγματι το 5, 10 ή 15 ή 30 90% του νερού που χρησιμοποιούμε προέρχεται μετά την ε, επεξεργασία και ανακύκλωσή του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ερμήνια Ματσόνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι επί της ουσίας ε, συμφωνούμε με το πόνημα του εισηγητή του κυρίου Ποστινάρου. Υπάρχουν προτάσεις που όπως είπα και σε προηγούμενες περιστάσεις υπάρχουν θέσεις στο κείμενό σας τις οποίες δεν ασπάζομαι. Όμως σε πλαίσια αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να θέσω τα εξή. Πιο συγκεκριμένα, κύριε Ποστινάρου, η θέση σας υπέρ της απομάκρυνσης, ε, αν θέλετε, η διεύρυνση των στόχων για τις επενδύσεις που μπορούν να δοθούν από Ταμείο Συνοχής. Και γενικότερα το που κάνει αυτή την πρόταση είναι κάτι που δεν συμμεριζόμαστε, γιατί οι ίδιοι στόχοι, όσο και αν γίνονται αποδεκτοί από όλους, μπορούν να καλυφθούν χρηματοδοτικά μέσω άλλων εργαλείων, χρηματοδοτικών εργαλείων. Είναι σημαντικό το σημείο εκείνο που αφορά την ρύθμιση της χρηματοδότησης από το Connecting Europe Facility. Πρέπει να υπάρξουν οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ε, στα πλαίσια του κανονισμού για το Ταμείο Συνοχής. Σας καλώ λοιπόν να το σκεφτείτε και πάλι, φυσικά και θα υποβάλω και μια σχετική τροπολογία. Θα σας υποβάλω μια τροπολογία καλώντας σας να αφήσετε ανοιχτό ένα παράθυρο για περαιτέρω τροποποίηση της πρότασης της Κομισιόν. Ζητώντας συγκεκριμένα ότι αυτοί οι πόροι θα πρέπει να μπουν στον εθνικό φάκελο στο μέτρο του δυνατού. Πολλές φορές έχω επίσης τοποθετηθεί σχετικά με το θέμα που προτείνει η Κομισιόν στο Γενικό Κανονισμό, όπου μεταξύ άλλων όρων να θέσει ως προϋπόθεση την μακροοικονομική προϋπόθεση. Με βάση την εμπειρία που έχουμε από τις χώρες παραλήπτες, αποδέκτες των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής. Και εδώ λοιπόν θα υποβάλω μια τροπολογία για το γενικό κανονισμό με σκοπό την απαλυφή αυτής της πρόβλεψης για μακροοικονομική προϋπόθεση και για το Ταμείο Συνοχής. Έχουμε και πρόσφατα πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούν χώρες που ήταν αντικείμενο στην εφαρμογή της ε, γιατί δεν είχαν τηρήσει αυτές τις παραμέτρους προϋποθέσεις που συνδέονται με αυτή την ερεσιμότητα, με αυτή τη συμμόρφωση και αυτές οι κυρώσεις οδήγησαν σε καταστροφικά αποτελέσματα για τις χώρες αυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η προϋπόθεση θα πρέπει να διαγραφεί. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι κάνοντας αυτή την πρόταση η Κομισιόν κάνει ένα βήμα πίσω. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η μακροοικονομική ε, πολλαπλή συμμόρφωση να απαλληφθεί από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι γενικότερα η στάση της Κομισιόν προσαρμόζεται στις παρούσες ανάγκες, παρούσες συνθήκες και επί της ουσίας σκόπιμο θα ήταν αυτή τη στιγμή να μην πιέζουν περαιτέρω, γιατί τους άλλους υπάρχουν γενικότερες ασάφειες και βεβαιότητες ε, σχετικά με την αναθεώρηση του προπολογισμού και γενικότερα ποια θα είναι η τύχη του Ταμείου Συνοχής και της Πολιτικής Συνοχής στη νέα προγραμματική περίοδο. Οπότε θεωρώ ότι με τις επιμέρους τροποποιήσεις που ζητούμε μπορούμε γενικότερα να στηρίξουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ήθελα επί της ουσίας να θίξουμε και να ζητήσουμε άρδιν τροποποίηση της πρότασης της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε άλλους δύο ομιλητές συν την Κομισιόν. Και κλείνω τον κατάλογο. Θα δώσω στους δύο ομιλητές 1,5 λεπτό στον καθένα. Ο Λάμπερτ Φανίστλερο είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σχόλια. Αν μπορώ να την αποκαλέσω έτσι, η ενεργειακή επανάσταση είναι κάτι το οποίο ξεκινά τώρα και θεωρείται σημαντικός στόχος. Θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε και στα κονδύλια συνοχής. Και γενικώ αν δει κανεί ε, και πέραν των διαδοτικών ταμείων, εκεί που θα ε, έχει μεγάλη σημασία για την μετάβαση, για την ενεργειακή μετάβαση, θα είναι το Ταμείο Συνοχής. Χθε συζητούσαμε για έλλειψη προθυμίας, ε, σίγουρα χρειάζεται και προθυμία και βούλης και διάθεση, αλλά το Ταμείο Συνοχής είναι μείζον. και θα μπορούσαμε να πετύχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Αν δει κανείς, παραδείγματος χάρη, τη μείωση εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα. Πρέπει να επικεντρωθούμε πρακτικά σε αυτά τα ζητήματα, παρότι είναι σημαντική στόχη. Πρέπει να φροντίσουμε και τα λεγόμενα revolving funds, τι θα γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να τα χρηματοδοτήσουμε όλα, χρηματοδοτούμε τη διαδικασία και μετά γίνεται από μόνο του το πράγμα κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι έχουμε και κατάντι πολλά ωφέλη στη συνέχεια τα οποία προκύπτουν. Και νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος που θα το στήριζε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την μακροαιρεσιμότητα, στο γενικό κανονισμό Λέμε ότι δεν είμαστε υπέρ. Αλλά θα έπρεπε να δούμε την ε, σημερινή κατάσταση. Παραδείγματο χάρη, τι λέει ο κανονισμό ε, για το Ταμείο Συνοχή σήμερα. Χρειάζονται και γι' αυτό χρήματα. Άρα πρέπει να έχουμε υπόψη μα και τι ε, σημερινέ πραγματικότητε. Δηλαδή πρέπει να διαχειριστούμε τα πράγματα κατά τρόπο ώστε να είμαστε συνεπείς. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας, αλλά όχι να υπερβούμε αυτά που κάνουμε, να ολοκληρώσουμε, να οριστικοποιήσουμε αυτά που κάνουμε. Και η έκθεση νομίζω όταν ολοκληρωθεί θα είναι πάρα πολύ καλή και θα μπορούμε να τη θέσουμε σε ψηφοφορία. Ναι. Και... Τώρα ο κύριο Τσέλερ, παρακαλώ πολύ στόμα. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πουστινάρο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση. Η αιρεσιμότητα, η μακροοικονομική, συμφωνούμε, δεν θέλουμε να προχωρήσει. Ωστόσο, στα θέματα της ενέργειας έχουμε το ερώτημα το εξή. Ότι η συζήτηση τώρα θα πρέπει να μας δώσει απαντήσεις για το πού καταρχάς θα κινηθούμε, γιατί έχουμε τον κεντρικό στόχο της παραγωγής ανάπτυξης, που σημαίνει καταπολέμηση της κρίσης, και πολλοί είναι πολιτικοί στα κράτη-μέλη οι οποίοι αναφέρονται στα αντιδιαρθρωτικά ταμεία λέγοντας ότι θα πρέπει να παραγάγουν ε, ανάπτυξη. Είναι βέβαια από τον οικονομικό τόκο το πιο μεγάλο στο πλαίσιο της ε, πολιτικής ε, συνοχής και διευθυντικής πολιτικής. Άρα λοιπόν, εάν προσδιορίσουμε μέτρα σχετικά με την ενέργεια, δεν θα πρέπει να είναι μέτρα ενεργητικά που προάγουν και την ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε αυτό το συνδυασμό. Επίσης, στην πολιτική συνοχής θα έλεγα ότι έχουμε να κάνουμε μια προσέγγιση η οποία στόχο έχει να στηρίξει τις πιο αδύναμες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους επιτρέψει να ανέβουν στο τρένο και να ακολουθήσουν και τις πιο προχωρημένες. Αλλά αυτό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό αναπερίπτωση και αναπεριφέρεια. Μπορεί να χρειάζονται υποδομές, μπορεί να χρειάζονται ε, όμως ε, και άλλα μέτρα, όπως μέτρα εργασία, ε, θέσεων εργασίας, απασχόληση δηλαδή, ή μέτρα κατάρτισης ή κάτι διαφορετικό. Επίσης, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπεται η ε, ως όριο ένα 2% για την ε, μεταβαση των ποσών αυτών από τα κράτη. Επομένως αυτό μειώνει ουσιαστικά το συνολικό όγκο των ε, διαρθρωτικών των ποσών που έρχονται από το διαρθρωτικό ταμείο και ουσιαστικά περιορισμό ακόμη περιστολή του ΑΕΠ. Θα έχει ίσως και δημοσιονομικές επιπτώσεις Γενικότερα και γι' αυτό όπως προβλέπεται στο δημοσιονομικό κανονισμό, το capping αυτό, το, το, το όριο δηλαδή του 2%, δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά την άποψή μου. Η Πρόεδρος, αγαπητοί φίλοι, έχουμε σοβαρό πρόβλημα χρόνου. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να παρατείνω την ημέρα, να εξασφαλίσω περισσότερες ώρες την ημέρα. Έχουμε όμως πολλούς ομιλητές και άλλα θέματα ακόμα. Σας δίνω ένα λεπτάκι να μιλήσετε, αλλά παρακαλώ όποιο. Ε, ξεπερνάει το χρόνο του να έχει υπόψη του ότι έχει ροκανίσει το χρόνο των άλλων συναδέλφων. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου, κύριο Βλάσακ, για την προσέγγιση του κυρίου Ποστινάρου. Ο λίγες μόνο παρατηρήσεις. Η εστίαση στην αποτελεσματικότητα, στην ενέργεια είναι πολύ σημαντική. Εγώ θα μιλούσα ωστόσο και για ευφυή δίκτυα και ευφυή ε, κτίρια που θα πρέπει να ενσωματωθούν σαν ε, όροι μέσα στις ιδέες αυτές. Στο διάρθρο 3 θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη σημασία μέτρων ε, καταπολέμησης πλημμυρών και συγκέντρωσης υδάτων, ομβρίων υδάτων. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενσωματωθεί και αυτό. Ευχαριστώ, Μαρτίν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. καθώ είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τι θέσει μα και στο παρελθόν. Ε, ιδιαίτερη εκτίμηση τρέφουμε καταρχά για την ε, δουλειά του εισηγητού, είναι εξαιρετική δουλειά. Είχαμε πολύ καλή επαφή σε όλο αυτό το διάστημα, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα προ τι προτάσει του. Ένα μόνο ερώτημα θα ήθελα να υπογραμμίσω. Ο συσχετισμό μεταξύ Ταμείου συνοχή ε, και του Connecting Europe του μέσου Connecting Europe, συνοδεύοντας την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ε, στον κανονισμό των κοινών προϋποθέσεων και δει στο 18.4, άρθρο 18, 4, υπάρχουν κάποιοι όροι και δεν νομίζω ότι, υπάρχει, ότι θα ήταν εύστοχο να αναπτύξουμε διαφορετικές διατάξεις σε διαφορετικά νομοθετήματα, δηλαδή στο κανονισμό το Ταμείο Συνοχή, στο Connecting Europe και το καθεξής. Στο... Γι' αυτό λοιπόν προτείνουμε εμείς και επιμένουμε ότι θα πρέπει να είναι στις γενικές διατάξεις σχετική όρη. Για δε την ουσία θα ήθελα να πω ότι ακόμη εξελίσσεται ο διάλογος ε, και η αναζήτηση της ορθής τη λεπτή αυτή ισορροπία που θα δοθούν οι προτεραιότητε, αλλά ασφαλώ μπορούμε και να ενσωματώσουμε στην νομοθεσία μηχανισμού ε, που να επιτρέπουν ε, την ευθυγράμμιση να χρειάζεται. Ξέρουμε ότι δεν συμφων... Ξέρετε ότι δεν συμφωνούμε να ε, επεκταθεί το θέμα της ενέργειας και της θερμότητας καλύτερα στην ιδιωτική στέγη. Ο Επίτροπος έχει δώσει τα επιχειρηματά του. Έχουμε μελετήσει πολύ προσεκτικά την υπόθεση αυτή και επιμένουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει το Ταμείο συνοχή να περιοριστεί στους κύριους στόχου του, στην κύρια στοχοθέτησή του και όχι να επεκταθεί. Ε, ο στόχο του περιορισμού των ε, εκπομπών είναι προφανώς διαρκή στόχο και δεν κάνουμε τίποτε που θα μπορούσε να υπονομεύσει το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών, τη σχετική συμφωνία και άρα περιορίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με ε, την παραγωγή κάτω από 20 ΜΒ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, θεωρεί ότι είναι καλύτερη μια οριζόντια προσέγγιση. Η σημασία της προσβασιμότητας είναι πολύ σημαντική, η προσβασιμότητα στις υποδομές που θα οικοδομούνται, θα κατασκευάζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά και πάλι μέσω των γενικών διατάξεων, μέσω των γενικών αρχών, όσον αφορά την ε, αρχή διαχείρισης αλλά και, όσο, και με την αιρεσιμότητα που προβλέπεται ε, σε συνδυασμό με την Σύμβαση των Ηνωμένων Αθηνών για άτομα με αναπηρίες νομίζω ότι καλύπτονται οι ανάγκες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επαναληφθούν οι ίδιοι όροι και διατάξεις εδώ μέσα γιατί μια επανάληψη διατάξεων που ήδη ισχύουν και αυτονόητα εφαρμόζονται θα οδηγούσε σε λάθος εφαρμογή. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τους συναδέλφους ε, για τα σχόλιά τους. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο από τους Πρασίνους σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα δώσω μεγάλη προσοχή στις ιδέες ε, που διατυπώσατε. Για την κυρία Ματσόνη, ο γενικός κανονισμός είναι ο χώρος όπου συζητούμε τα θέματα της μακροοικονομικής ερεσιμότητας. Εγώ είμαι Αντίθετο, κάθετα αντίθετο με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Εξού και έχω καταθέσει και σχετική τροπολογία, αλλά για τον γενικό κανονισμό. Γιατί στην δική μου έκθεση δεν είναι ο κατάλληλο χώρο για να εξετάσουμε τα ζητήματα αυτά. Δεν θέλω δηλαδή να μπω σε τομεί ε, ή σε χωράφια, αν θέλετε, των ε, συνεισηγητών, των, των φίλων για τον γενικό κανονισμό. Διεύνηση τώρα του πεδίου εφαρμογή ε, του Ταμείου Συνοχή. Το πρόβλημά μα ποιο είναι. Να λύσουμε προβλήματα που δεν είναι απλά πραγματικά, αλλά ορισμένες φορές είναι και δραματικά. Και σίγουρα πολύ μεγάλο θέμα εξοικονόμηση ενέργεια ε, για τις κατοικίες, μείωση εκπομπών δεξιδιού του άνθρακα, βελτίωση ενεργειακού μείγματος. Όλα αυτά είναι αναγκαία. Και πολλές φορές το έχει πει και η Επιτροπή των Περιφερειών. Και το Συμβούλιο το έχει πει, το ξέρει η Κομισιόν. Επίσης πολλοί συνάδελφοι και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μας ε, το έχουν πει. Και απευθύνομαι κυρίως στον συντονιστή του ΕΛΚ ε, Φανίστερο και τον ευχαριστώ που στηρίζει αυτή την πρόταση. Τώρα για τον κύριο Τσέλερ. Πράγματι, ένας βασικός στόχος ε, του Ταμείου Συνοχής είναι η μείωση των ανισοτήτων του χάσματος που υπάρχει μεταξύ περιφερειών και εντός περιφερειών. Αν χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Συνοχή ε, για την εξοικονόμηση ενέργεια, για τη δημιουργία τοπικών πράσινων θέσεων εργασία και τη δημιουργία καλών συνθηκών διαβίωση για του πολίτε μα, για τη δημιουργία χώρων ε, λιγότερο ε, μολυσμένων, με μικρότερη ρήπανση, είναι ένα καλό τρόπο για την καταπολέμηση αυτών των ανισοτήτων. Εξού και το προτείνω για την εκπαίδευση και κατάρτιση, κυρίως εδώ μπαίνει το κοινωνικό ταμείο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να μπει και το ταμείο συνοχής. Για τα εφή κτίρια, τα έξυπνα κτίρια, το λέω και στην έκθεσή μου, ε, δεν το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα χρησιμοποιήσω την ε, δική σας έκφραση για να το πούμε πιο ρητά και να εξηγήσουμε τη φιλοσοφία μας καλύτερα. Και για την... Ε, αντιπλημμυρική προστασία και αυτό είναι μια καλή ιδέα και θα την ε, εντάξω. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέσο για το Connecting Europe, η Κομισιόν δεν είναι υπέρ να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε μνήμα στον τρόπο με τον οποίο θα μεταφέρονται οι πόροι και υπό ποιες προϋποθέσεις. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει σαφής αντίδραση από ορισμένα κράτη-μέλη που είναι αντίθετα στη σημερινή φιλοσοφία του Connecting Euro. Πρέπει να έχουμε πίσω την πραγματικότητα. Εάν θέλουμε να είναι βιώσιμο, να είναι πραγματικό αυτό το έργο, να φέρει αποτελέσματα, και εγώ είμαι υπέρ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις ανησυχίες που υπάρχουν, όχι μόνο εντός ε, Συμβουλίου, αλλά και εδώ στην Επιτροπή μας. Εξού και έχω καταθέσει αυτή την τροπολογία, διότι τελικά Πρόκειται για τη μεταφορά 10 δι ευρώ από το Ταμείο συνοχή. Δεν θα πέσουν από τον ουρανό αυτά τα χρήματα και δεν βλέπω κάποιον συνάδελφο από την Επιτροπή Ρέγγι ε, να θέλει να το πράξει αυτό χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση. Εγώ θέλω να υπάρχουν εγγύησεις, να υπάρχουν όροι, προϋποθέσεις. Γι' αυτό και συνεργάστηκα πολύ στενά με την ΓΔ Ρέγγιο Είχα επαφέ και με την Επιτροπή των Περιφέρων και με τη ΓΔ Ρέγκιο τη Κομισιόν. Ζήτησα από του δύο επιτρόπου, τον Κάλλα και τον Χαν, να υποβάλουν μια κοινή πρόταση. Τώρα, πότε αυτή η πρόταση θα είναι έτοιμη, θα δούμε. Θα είμαστε κι εμεί ε, έτοιμοι τουλάχιστον να το μελετήσουμε και να το εντάξουμε στην δική μα έκθεση. Σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργεια είναι κάπω επιφυλακτική η Κομισιόν από ό,τι βλέπω. Παρουσιάζει κάποιε ενστάσει. ελπίζω όμω το τέλο να επικρατήσει αυτή η φιλοσοφία. Δεν έχει να κάνει με τη δική μου έκθεση, ξέρετε. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι πρέπει να γίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ζητά να γίνει το Συμβούλιο. Και πολλοί επιτρόποι είναι υπέρ και το στηρίζουν και πολλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές. Τέλος, προσβασιμότητα. Ναι, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι οι δικές μου τροπολογίες ε, κάπως αλληλεπικαλύπτονται με το γενικό κανονισμό. Αν είναι έτσι όμως, γιατί με κυβερνητικέ οργανώσεις αγωνίζονται, παλεύουν για τα άτομα των ανθρώπων με αναπηρία. αφού έχουν μπει τα σχετικά στους οριζόντιους κανονισμούς, δεν είναι κακό. Εμείς θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι περιλαμβάνει ο γενικός κανονισμός θα ενσωματωθεί και στις οριζόντιες εκθέσεις μας. Όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με τους ειδικού αναταμιοκανονισμούς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ναι καταλαβαίνω για τα νομοθετικά αυτά ζητήματα σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι αύριο έξω το απόγευμα λίγη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη έκθεση. Δυστυχώς ε, έχουμε μείνει πίσω κατά ένα τέταρτο, άρα θα πρέπει να κόψω το χρόνο που θα δώσω για την ε, κάθε μία της επόμενης εκθέσει κατά τρία λεπτά. Επόμενη λοιπόν έκθεση, η έκθεση της κυρίας Ρίκα Μάνερ. Όσο θα μιλάει η κυρία Μάντερ, παρακαλώ να σηκώνετε το χέρι θέλετε να λάβετε το λόγο, γιατί μόλις ολοκληρώσει την παρουσίασή της κυρία Μάντερ θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Ρίκα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας πω ότι για την έκθεση αυτή έχουμε συμφωνήσει με τους συναδέλφους στα πιο πολλά σημεία. και δεν έχουν γίνει από την τελευταία φορά που συνεδριάσαμε ουσιαστικές αλλαγές. Θέλω να αναφερθώ στα μείζωνα ζητήματα, πρώτα απ' όλα για τον προπολογισμό, θέλω να πω λίγα λόγια. Είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει με τους κοιόδες ιδιαίτερα και θεωρώ ότι ως εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου θα πρέπει να κρατήσουμε τη γραμμή του 7% για τις κοινέ διατάξεις. Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό, τα πράγματα μας περιορίζουν πολύ ε, βάσει το πλαισίου που υπάρχει και το 3% ε, που προτείνει η Κομισιόν τελικά δεν θα παραμείνει, ε, θα πέσει κάτω από αυτό, γι' αυτό θα πρέπει να εμείνουμε στο 7% από πλευρά μας όσοι ε, είσαστε προσπάθεια να ε, υπερασπιστούμε τελικά και να καταφέρουμε να επιτύχουμε 3% της πρότασης της Κομισιόν σε ό,τι αφορά τώρα τις προτεραιότητες επενδύσεων. Αν επιθυμούν οι συνάδελφοι να υποβάλουν τροπολογίες, παρακαλώ να λάβετε πόσο κατά πόσο τροπολογίε ε, που υποβάλλετε κινούνται προ την κατεύθυνση των προτεραιοτήτων του Ταμείου του Περιφερειακού και κατά πόσον ε, συνάδουν και με ε, το, τα προγράμματα ETC. Ε και θα έχουμε συνεργασία με τον η συγητή αρμόδιο για τις προτεραιότητες ε, του Περιφερειακού Ταμείου, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε πιο συντονισμένα. Πιστεύω ότι ο στόχος είναι να στηρίξουμε την περιφερειακή συνεργασία και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τα σχετικά κονδύλια. Άλλοι τώρα τομείς, άλλα πεδία ενδιαφέροντος να πω ότι η χρηματοδότηση ETC φτάνει το 150% η στήριξη λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Δεν ξέρω τελικά τα επίπεδα αυτά δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν στο τέλος δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε απόλυτοι στα αριθμητικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τα καταπληκτικά, ποσά, βλέπετε ότι εγώ προτείνω 20% αντί 15%. Αν τελικά τα βασικά προγράμματα προσαρμοστούν στο 20% τότε θα τροποποιήσω την πρότασή μου. Αναλόγως. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, την Ευρωπαϊκή Εθνική Συνεργασία να προτείνουμε ένα καταποκοπήν ποσοστό 5-10% υψηλότερο. Σε ό,τι αφορά την ευελιξία ανάμεσα στις διάφορες συνιστώσεις α και β, 15% είναι το ποσοστό που θα προτείνουμε θέλουμε να διαφυλάξουμε την ευελιξία και στην επόμενη προγραμματική περίοδο και υπήρξε συμφωνία με τους ισχυώδεις επ' αυτού. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θεματική συγκέντρωση, υπήρξε ουσιαστική συμφωνία ανάμεσα στους αδέλφους και με τους ε, Εγώ προτείνω ε, πέντε θεματικές ενότητες και όχι τέσσερις. Υπάρχει λοιπόν μια συμφωνία και από αυτό. Αν δούμε τώρα τους δείκτες, θα δούμε είναι ένα θέμα που μας απασχόλησε τελευταία συνεδρία. Ο συνάδελφος ε, Πόστα και το δικό του κείμενο γίνεται κάποιες αντιπροτάσεις. Στο δικό μου κείμενο τελικά προτείνω ότι οι τελικοί αυτοί δείκτες καλό είναι να μεταφερθούν στην κατεξιοδότηση πράξης. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση πρόγραμμα είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει στο τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα και Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι θα υποβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση τροπολογίες. Σε παλαιότερη έκθεση ε, είχε θίγει το ίδιο ζήτημα και μετά από τις διαπραγματεύσει που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης ένα πρόγραμμα είναι κάτι που δεν ε, αλλάζει ω στρατηγική και δεν θεωρώ ότι είναι καλό να κάνουμε τέτοιου είδου αντιπροτέ αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ ε, και πάλι για την καλή συνεργασία. Ε, ελπίζω να έχετε να κάνετε και άλλε καλέ προτάσει και τροπολογίες ε, στην έκθεσή μου. Ο πρόεδρο. δεν θέλει να μιλήσει πέρα από του σκιώδεις, οπότε κλείνω τον κατάλογο. Τέσσερι σκιώδεις έχουν το λόγο. Λαμπέρ και ρωτώ ποιοι, ποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Εσείς είστε σκιώδες, σας έχω συνυπολογίσει. Άρα μόνο Λαμπέρ. Έναν ε, ομιλητή λοιπόν έχω και τέσσερις σκιώδες, τρία λεπτά για κάθε σκιώδη. Ο κύριος Διάντζελης ε, πρώτα απ' όλα. Τρία λεπτά. Ε, Ευχαριστώ. Είμαι της γνώμης ότι πραγματικά είναι αξιέπαινη η δουλειά που έκανε η συγγήτρια και σε ό,τι αφορά την δεύτερη σειρά των τροπολογιών και θα μπορούσα να πω ότι έχει πετύχει απόλυτα το στόχο της, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά μια πιο φιλόδοξη εδαφική συνεργασία και μια πιο εύρωστη, αν θέλετε, ε, εδαφική συνεργασία. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και την κατανομή των κονδυλίων, σε ό,τι αφορά την εδαφική ε, συνεργασία, αναμφίβολα, ε, ο στόχος του 7% είναι πολύ φιλόδοξος. Στο παρελθόν αυτό έχει επιβεβαιωθεί και εδώ στο Κοινοβούλιο αναφέρομαι στην έκθεση Σάντσεθ Σμιθ. Στο μεσοδιάστημα Βεβαίως έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στην Ευρώπη, ιδίως σε ό,τι αφορά συνολικά την πολιτική συνοχή. Δυστυχώς, η πρόταση αυτή τη στιγμή που είναι στο τραπέζι κινείται πολύ χαμηλότερα από ό,τι προβλέπει η παρούσα προγραμματική περίοδος, οπότε ένα αίτημα πλευράς Κοινοβουλίου που φτάνει το 7% ουσιαστικά θα σημαίνει να γίνει αποδεκτός μείωση άλλων σημαντικών κονδυλίων από άλλους ε, τομείς της πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει λοιπόν ναι μεν να ενισχύσουμε το διαπραγματευτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και αναμφίβολα ο στόχος του 7% αν μην σε αυτόν μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Όπως πολύ ορθά είπε και η συγγήτρια ίσως αν εμείνουμε ε, σε αυτό το 7% διαπραγματευτικό χαρτί, να καταφέρουμε τελικά να κρατήσουμε το 3% που προτείνει η Κομισιόν. Στα υπόλοιπα ζητήματα τώρα, ε, συμφωνώ με όλα όσα αφορούν την ευελιξία. Όπως και σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση. Ιδίως ε, σε ό,τι απαιτείται των στόχων. Μπορώ να ανοίξω μόνο μια παρένθεση για τρία ζητήματα που θεωρώ μείζονο σημασία σε ό,τι αφορά την χρήση των διευθυντικών ταμείων, τα οποία είναι τα εξή. Απλούστευση και μεγαλύτερη ευελιξία. Κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου για την διευκόλυνση στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση πιστεύω ότι όλοι είμαστε υπέρ της βελτίωσης της προσβασιμότητας της χρηματοδότησης. Έχουμε να κάνουμε σημαντικά κονδύλια, σημαντικούς πόρους, ιδίως σε μια τόσο δυσχερή ε, συγκυρία και σε μια τόσο έντονη ε, κρίση λοιπόν. Άρα ευελιξία, απλούστευση, άρση της γραφειοκρατίας. Δεύτερο και σημαντικό ζήτημα κατά με είναι το ζήτημα των προτεραιοτήτων αλλά και η ποιότητα των στόχων επί των οποίων επενδύουμε. Η ποσότητα ναι μεν είναι σημαντική, αλλά πιο πολύ σημαντική είναι η βέλτιστη χρήση των πόρων, άρα η ποιότητα των στόχων, η ποιότητα των project που θα τύχουν ε, χρηματοδότησης. Η, η χρηστή χρήση των πόρων ε, εν τέλει αν θέλετε και ε, είμαι της γνώμης ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις που έχουν γίνει και στα πλαίσια της διάσκεψης των Πρόεδρων υπήρξε μια συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων ότι η κοινοβουλευτική δραστηριότητα δεν πρέπει να κινηθεί ενάντια την ισορροπία του προπολογισμού. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο και περίπλοκο ζήτημα αυτό. Θέλω να σταματήσω εδώ. Θέλω να επαναλάβω ότι η δουλειά που έκανε στη γήτρια είναι εξαιρετική πολύ, ε, και πολύ θετική. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Φρανσουά Αλφόνση, παρακαλώ, επενθυμίζω, μην υπερβαίνετε το χρόνο σας, γιατί τελικά δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την τελευταία έκθεση. Θα προσπαθήσω, κυρία Πρόεδρε, να κάνω αυτή την προσπάθεια. Θέλω να πω στην εισηγήτρια ότι συμφωνούμε με την ουσία των προτάσεών της και ιδίως με την φιλοδοξία σε ό,τι αφορά το στόχο του 7% για τα κονδύλια που πηγαίνουν προς την εδαφική συνεργασία και σε ό,τι αφορά την ευελιξία επίσης για τη συμπερίληψη των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος στους στόχους και στις επιλέξιμες υπηρεσίες και στις παρεμβάσεις της εδαφικής συνεργασίας και συμφωνούμε και με την διεύρυνση της, εδαφικής, της, συγγνώμη, της θεματικής συγκέντρωσης γύρω από πέντε θέματα και όχι τέσσερα. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω, τα οποία μας δημιουργούν κάποιες ανησυχίες. Πρώτα απ' όλα τα νησιά. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε ε, μια κατάσταση που ίσως είναι ιδιαίτερη, αλλά υπάρχουν κάποια κριτήρια ε, των 105 χιλιόμετρων και ε, το νουτς 3, αυτό το κριτήριο. Ένα νησί δεν είναι ένα σύνορο όπως σε ένα χερσαίο σύνορο. Πρέπει να περάσει κανείς από ένα λιμάνι, από ένα αερολιμένα που μπορεί να είναι σε ένα ή άλλο νομό της, ε, του νησιού αυτού. Και εκεί υπάρχει εμπλοκή ε, στα προγράμματα. Αν πούμε παραδείγματο χάρη ότι με την Τινησία μπορεί να συνεργαστεί μόνο η Νότια Σικελία ή ξέρω εγώ ε, με κάποια άλλη χώρα, η Κορσική μόνο το βόρειο τμήμα κτλ. Αυτό το κριτήριο των 150 χιλιόμετρων δεν επιτρέπει παραδείγματο χάρη στην Κορσική να έχει συνεργασία με τις Βαλεαρίδες ενώ υπάρχουν τουριστικές, περιβαλλοντικές δραστηριότητες που καλούμαστε να έχουμε συνεργασία και δεν μπορούμε. Άρα, καλό είναι να υπάρξει ίσως όχι παρέκκληση ως προς την αρχή, αλλά ως προς την πρακτική εφαρμογή, γιατί ε, το νησί είναι ένα σημείο εισόδου. Θέλω να καταλάβουν οι συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντικό για τις νησιωτικές περιοχές. Θέλουμε να συμμετέχουμε στην εδαφική ε, συνεργασία Είμαστε και ένα σημείο διασύνδεσης ε, των ε, διαφόρων ε, περιφερειών και λεκανών. Δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι υπάρχουν κάποιες κοινές κάποια κοινά πολιτιστικά στοιχεία σε όμορες περιοχές. Ε, κοινέ κουλτούρε αν θέλετε. Αυτά πρέπει να τα προβάλλουμε αυτά τα στοιχεία για να τονίσουμε την ένωση ε, που υπάρχει ε, στην Ευρώπη. Να μην προβάλλουμε τι διαφορέ διαφορές αλλά και τα σημεία που ενώνουν. Ο κύριο Βλάσεκ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λίγα σχόλια. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η χρηματοοικονομική πόρη, το 7% είναι υπερβολικά φιλόδοξο κατ' εμέ. Με το 3,5% θα ήμουν ικανοποιημένο. Αυτό που προτείνεται δηλαδή. Τώρα, προτεραιότητες στις επενδύσεις. Νομίζω ότι για την διασυνορική συνεργασία Πολύ σημαντικό είναι να βελτιωθούν ε, οι υποδομές που δεν είναι καλές, ε, να μην έχουμε συμφορήσεις ε, στα δικτυά συγκοινωνιών μεταφορών και κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να στηρίξουμε είναι οι πολιτισμικές ανταλλαγές και βελτιωτικών υποδομών. Που είναι μια καλή πηγή για εξέβρεση θέσεων εργασίας. Θέλετε το λόγο. Κυρία Μάλση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μία παρατήρηση γενικής φύσεως για να συμφωνήσω με αυτά που έλεγε στον Αλφος για τις ε, άκρως κέντρες περιφέρειες που κυρίως ε, είναι νησιωτικές περιοχές. Το ζήτημα της αταφικής συνεργασίας είναι θεμελιώδες για τις περιοχές αυτές. Αληθεύει ότι το κριτήριο των 150 χιλιόμετρων πολύ συχνά δημιουργεί προβλήματα. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι οι από απόκεντρες περιφέρειες αυτές είναι σε επαφή και με χώρες ΑΚΕ, δηλαδή από, τις, ε, από την Αφρική, την Καρευκή και τον Ειρηνικό. Και σε θέματα συνεργασίας σίγουρα αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα ή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ε, έχει κοινέ αξίες, ε, ιδίως πολιτιστικές, πολιτισμικές αξίες με τις χώρες αυτές. Και μπορούν έτσι να διαδοθούν αυτές οι αρχές, οι κοινέ. Δεύτερη παρατήρηση για τη ε, διασυνοριακή συνεργασία. Νομίζω ότι και εδώ συμφωνώ με αυτό που ήθελε να πει ο Σεναλφος Αλφονσί. Θεωρώ ότι οι περιφερειακές γλώσσες έχουν μεγάλη σημασία. Πρέπει να τις προβάλλουμε. Περιφερειακές γλώσσες που ε, είναι και διαδεδομένες στη λεκάνη με την οποία είμαστε σε επαφή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λάμπερτ. Thank you very much. Just a couple of, of, of remarks. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ τις παρατηρήσεις. Είναι σοφό πιστεύω να έχουμε μια σειρά από διατάξεις για την εδαφική συνεργασία ώστε να έχει τη σωστή θέση και να ενισχυθεί ακόμη η θέση του τι μπορούμε να κάνουμε με εδαφική συνεργασία υπερσυνοριακή, διαπεριφερειακή μεταξύ χωρών. Και θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε την διάσταση της μακροπεριφερειακής συνεργασίας και να την εντάξουμε στην εδαφική συνεργασία με άξονα δηλαδή την εδαφική συνεργασία στην πολιτική συνοχή. Και έτσι με τον τρόπο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω το πού μπορούμε να το εντάξουμε είχαμε την ακρόασή μας αυτές με διαφόρους ερευνητές, με διαφόρους φορείς και εκπροσώπους που, που ε, δραστηριοποιούνται ε, και θα ήθελα να πω ότι μέσα στην πρόταση του ορίστου του 2020 ένα μεγάλο πρόγραμμα που ονομαζόταν Περιφέρειες της Γνώσης θα πρέπει να μεταφερθεί στην πολιτική συνοχής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να διαφυλάξουμε αυτή τη δυνατότητα. Και ιδιαίτερα, όταν μιλούμε για έρευνα και ανάπτυξη και πορεία για αριστεία, θα πρέπει στην εδαφική συνεργασία να, δώσουμε μια, να προσδώσουμε μια νέα διάσταση, που πιστεύω στα επόμενα 7 χρόνια πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί. Για το 7%. Το 7% στα συγκεκριμένα πλαίσια είναι επιλογή του Κοινοβουλίου. 7% που έχουμε ήδη συμπεριλάβει και σε άλλη έκθεση και στις συζητήσει μας για την περίοδο 2007-2013 είχα και συζητηθεί, αλλά απλώς τότε το Συμβούλιο οπισθοδρόμησε. Είχε μια πιο συντηρητική, μια πιο σφιχτή στάση, ενώ το Κοινοβούλιο ήταν πολύ πιο ε, φιλόδοξο και τους τραβήξαμε. Νομίζω λοιπόν πρέπει να επιμένουμε στην μακροπεριφερειακή διάσταση. Και επίσης να δούμε μια τελείως νέα ε, διάσταση στην περιφέρεια της γνώσης. Πώς θα ορίσουμε την περιφέρεια της γνώσης. Πρέπει νομίζω να την ε, υπογραμμίσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Σάμψη Σμιτ είναι στην αντιπροσωπεία της τώρα, γι' αυτό δεν μπορούσε να έρθει, αλλά πάντως ε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν από την Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ επικοδομητική συνεργασία στην έκθεση της. Υπάρχουν ε, πολλές καλές βάσεις ε, επαφής και ε, σύγκλησης πιστεύω στις προτάσεις αυτές. Πολλές από τις ε, προτάσεις διευκρινίζουν σημεία της διατύπωσης της προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό τις θεωρούμε χρήσιμες. Θα επικεντρωθώ σε τούτο μόνο σε κάποια σημεία στα οποία δεν είμαστε τόσο σύμφωνοι. Όσον αφορά την ε, κατανομή των ποσών των δημοσιονομικών πακέτων. Θα το δούμε βέβαια και με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το ETC ε ε, αποτελεί ένα χώρο προσθέμενης αξίας και θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη και τα πρακτικά ζήτηματα, αυτά που εκπείρας διαπιστώνουμε, ότι απαιτούν να λειτουργήσουν ε, τα ταμεία αλλά που ε, περιπλέκουν περισσότερο γιατί προστίθεται και μια επιπλέον διάσταση, δηλαδή η κρατική διάσταση. Αυτά λοιπόν θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ως προς τις προτάσεις ε, στον τομέα αυτών. Επίσης, ανησυχίες έχουμε επί της ουσίας στη θεματολογική συγκέντρωση και τα σχετικά σημεία. Πάλι είναι δύσκολο βέβαια να εξισορροπηθεί σωστά το σύνολο των προτάσεων. Στα προγράμματα έτσι έχουμε μια σειρά από διασυνοριακά προγράμματα με σημαντικούς, ε, σημαντικά ποσά για τη χρηματοδότηση. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ανοίξει το πεδίο των ε, τομέων που θα καλυφθούν έστω, αλλά δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει να αναμειχθούν διαφορετικά θέματα στην ε, κατά πρόσβαση. Αυτό έχει νόημα μόνο στην βασική ε, πρόσβαση στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη για του 11 δηλαδή στόχου. Αλλά όταν μιλούμε για συγκέντρωση μόνο σε ορισμένου θεματολογικού θεματικούς στόχου, δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε τόσο περίπλοκες ε, λύσεις και ως προς τη διαχείρισή τους. Γιατί βέβαια και η παρακολούθηση της χρηματοδότησης θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικούς ρυθμούς και σε διαφορετικό επίπεδο. Για τις προτεραιότητες, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε την εξή προσέγγιση. Ξεκίνησε με τις βασικές προτεραιότητες του κανονισμού, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και στη συνέχεια τους εμπλούτησε τους στόχους αυτούς Ε, κατά τρόπον ώστε να συνδυάσει με το ETC ε και να φτάσει στο συνδυασμένο ε, τύπο χρηματοδότηση που ονομάζουμε χρηματοδότηση ESF. Εδώ λοιπόν έχουμε ειδικές, ε, ιδιαίτερες προτεραιότητες χρηματοδότησης στο ETC που σε ορισμένες περιπτώσεις συμπίπτουν με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, φέρει ε, οικονομικές υπηρεσίε γενικού συμφέροντο. Όλα αυτά λοιπόν, δημοσίου συμφέροντος, όλα αυτά λοιπόν τα λέμε για να υπογραμμίσουμε ότι πρέπει πάντα οτιδήποτε το επιπλέον προτείνεται να είναι εστιασμένο και απαραίτητο. Γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό πάντοτε. Από άλλες συστήσεις επίσης θα γνωρίζετε ότι έχουμε πολλές επιφυλάξεις ως προς τη συμπερίληψη και του τουρισμού σαν ρητή διατύπωση ενός στόχου ανάπτυξης, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε ε, στόχο επένδυσης, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με ε, στόχους και όχι με στόχους ανάπτυξης, Επένδυση, συγγνώμη. Έτσι λοιπόν, θα ήταν ε, εσφαλμένο το μήνυμα το οποίο θα προστελόταν αν συμπεριλαμβανόταν ο, ο τουρισμός ως το κλάδος επενδύσεων σε ορισμένε περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να, προ... να προαχθεί, αλλά όχι εν προκειμένου. Επίσης θα πρέπει να δούμε στις ε, κανονιστικές προτάσεις, όπως είπε ο κ. Ρόι, ε, τι είδους ε, αποτύπωμα υπάρχει από τις προτάσεις σας. Για τις ε, τροπολογίες θα έλεγα ότι τα πράγματα έχουν ήδη καλυφθεί και θα ήταν καλό να εξετάσουμε προς τα που μπορούν να οδηγήσουν. Για τις ε, άκρες απομαξιμένες περιοχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ε, εγγύηση του 150% των πιστώσεων προκειμένου να έχουμε ε, εξασφαλισμένο ότι θα γίνεται κάτι συγκεκριμένο και εστιασμένο στις ε, άκρους απομακρυσμένες περιφέρειες. Μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω και να διερευνήσουμε ποιες είναι πράγματι οι ανάγκες του σε κάθε περίπτωση και η Επιτροπή βέβαια είναι αποφασισμένη να το πράξει και να το επιτύχει. Όσον αφορά τις σχέσεις με το ΕΠΑ και το ΕΑΝΑΕ, ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν και το βλέπουμε από την πείρα μας είναι ότι η χρηματοδότηση που δεν απορροφάται δεν θα πρέπει να πηγαίνει σε προγράμματα εξωτερικά, έξω, των, έξω από τα σύνορα δηλαδή. Υπάρχει λόγος που είναι περιορισμένα μόνο στην ενδοκινοτική, στην ευρωπαϊκή διάσταση μόνο. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα ήθελα να υπογραμμίσω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για του δείκτε είναι ότι πρέπει οι δείκτε να προσδιορίζονται προκαταβολικά, εξάντε. Και αυτό ισχύει για όλου του κανονισμού, για όλα τα προγράμματα. Για να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενο τι είδου ε, συστήματα ε, παρακολούθηση εποπτείας θα εφαρμόζονται, πώς θα μπορεί δηλαδή να είναι και ο ίδιος ε, ευθυγραμμισμένος με τους δείκτες αυτούς. Προκαταβολικά και να εξασφαλίζεται και η συνοχή των δικτών που χρησιμοποιούνται μεταξύ διαφόρων ταμείων, ώστε και η Επιτροπή από πλευρά της να μπορεί να ε, καταθέτει τις εκθέσεις της και να δίνει να αποδίδει λογαριασμό για τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο η εισηγήτρια παρακαλώ για να ολοκληρώσει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ επικοδομητικά σχόλια. Πολύ στόμα μόνο κάποιες παρατηρήσεις, ολίγες παρατηρήσεις. Για τον κύριο Ντεάντζελης, για την ε, απλούστευση. Νομίζω ότι έχει ήδη λάβει υπόψη τη διάσταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς λέγει ότι ενσωματώνονται στο πρόγραμμα οι έλεγχοι. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο. Επίσης, τα 150 χιλιόμετρα που έχουν συζητηθεί σε διάφορα επίπεδα και συστηθεί σε ένα δύσκολο θέμα θα ήθελα να υπογραμμίσω πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δίνει ένα περιθώριο διακριτικής ευχαίρειας με τις προτάσεις της. Και εδώ έχουμε να κάνουμε ένα όριο το οποίο αφορά μόνο τα υπερσυνοριακά ε, ε, προγράμματα. Τα διεθνικά προγράμματα έχουν διαφορετικούς όρους και μέσα σε διαφορετικό πλαίσιο θα αναπτυχθούν. Άρα νομίζω ότι μπορούμε με πολύ ε, επιτυχημένο τρόπο στο πλαίσιο αυτό να καλύψουμε το θέμα των θαλασσίων λεκανών, Φερρυπίν. καθώς το όριο αυτό των 150 χιλιόμετρων αφήνει πολύ μεγάλο περιθώριο ευχέρειας. Τα, ε, τα νησιά Φερρυπίν θα είχαν ε, μέσω των διευρωπαϊκών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων κάποιες, ε, κάποια υποστήριξη. Για τα σχόλια του κύριου Φλάσακ και τις προτεραιότητες. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τη γραμμή σας. Το πρόβλημα των στενοπών στην κυκλοφοριακή κίνηση λαμβάνεται υπόψη, πιστεύω και μπορούμε πολλά να επιτύχουμε, πολλά να βελτιώσουμε χάρη στην ε, διαπεριφερειακή συνεργασία. Για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, για τις ε, προτεραιότητες στην, στις επενδύσεις, θα ήθελα εξ αρχής να δηλώσω ότι θα προσπαθήσουμε μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης να εξασφαλίσουμε στόχους αποφεύγοντας τις επικαλύψεις. Για τον κύριο Φανίστηλ θα πρότεινα να συζητήσουμε ε, τις λεπτομέρειες διμερός ε, σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών προβλέπεται για αύριο στις 6 το απόγευμα. Παρακαλώ τώρα την κυρία Ιριγκόιεν Πέρες να κάνει την παρουσίαση της. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ήδη σας έχει διατεθεί η έκθεσή μου εδώ και κάποιες ημέρες σε όλες τις γλώσσες εργασίες, οπότε δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα σημεία. Απλά θέλω να προχωρήσω τη συζήτηση αναφερόμενη στις τροπολογίες που θα υποβάλω για να βελτιώσω περαιτέρω το κείμενο. Πρώτα απ' όλα μια τροπολογία σχετικά με την εφαρμογή της σημασίας που έχει η δημιουργία και η ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι πραγματική πηγή απασχόλησης. Δεύτερον, υποβάλλω κάποιες τροπολογίες επιμένοντας πόσο σημαντική είναι η διεθνική συνεργασία και θα πρέπει να λάβει υποχρεωτικά και όχι προαιρετικό χαρακτήρα και θα πρέπει να εφαρμόζεται πέρα από την κοινωνική κοινοτομία στους επιχειρησιακούς άξονες και επιχειρησιακά προγράμματα. Έπειτα έχουμε μία σειρά τροπολογιών στο παράδειγμα για τους δείκτες για να επισημάνουμε ότι όλα τα στοιχεία θα πρέπει να συγκεντρώνονται Αναφύλα για να γνωρίσουμε ακριβώς πώς κατανέμεται οι αν ανάμεσα στα φύλλα. Και θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με ε, τους δικιούς οικείχους που έχουν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα και καμία παροχή. Θα πρέπει έπειτα μεσοπρόθεσμα ακροπλασμά να ε, δούμε τι θα κάνουμε ακριβώς με αυτά τα άτομα που ε, έχουν μείνει χωρίς καμία στήριξη από το σύστημα πρόνοιας. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω θερμά τους σκιώδεις για την ουσιαστική τους υποστήριξη ε, στην έκθεση αυτή και την αποδοχή των τροπολογιών. Ξέρετε ότι η υποβολή τροπολογιών γίνεται μέχρι αύριο και 20 και 21 του μηνός θα συζητηθεί ε, και θα υπάρξει οφορία για το θέμα. Λοιπόν, περιμένω από τη σημερινή συζήτηση να ακούσω περαιτέρω σκέψη και ιδέες. Σας ευχαριστώ. Ε, ε? Θέλει κανείς το λόγο πέρα από τους κοιόδης. Κάποιος άλλος προς τους ε, Ξεκινάμε από το σκιώδη του ΕΛΚΑ, την κυρία Ζεύκα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι ένα θέμα αυτό που συζητούμε για πολλωστή φορά. Έχουμε ήδη θέσει προτάσεις Έχουμε ήδη υποβάλει που αποδέχθηκε η συγγήτρια και έχει εντάξει στο κύριο σώμα τη εκθεσή τη. Θεωρώ ότι η έκθεση ε, κινείται σωστή κατεύθυνση. Μιλά πλέον για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ω την ραχοκοκαλιά τη οικονομία και ότι είναι υπεύθυνε για την δημιουργία των θέσεων εργασία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή τη διατύπωση. Ε, ήταν κάτι που έλειπε αρχικά σε αυτή την έκθεση και από πλευρά μου θα ήθελα να αναφέρω και το εξή μιλήσατε ε, για τον ε, διεθνικό χαρακτήρα της ε, συνεργασίας και το ότι θα πρέπει να λάβει υποχρεωτική μορφή αυτή η συνεργασία, να μην είναι πλέον προαιρετική. Η διεθνική, αν θέλετε καλύτερα διαπεριφερειακή, θα προτιμούσα να πω, συνεργασία είναι κάτι σημαντικό. Στις δικές σας τροπολογίες, κυρία Σύγετρια μιλάτε και για τις ε, πιο ηλικιωμένες ηλικιακές μονάδες, ε, ε ομάδες συγγνώμη, πληθυσμού. Ε, θα κάνω μια τροπολογία ακριβώς για αυτόν τον όρο. Καλό να μιλήσουμε για τις ηλικίες 50 συν. και για τον ευάλωτο χαρακτήρα που έχουν ηλικίες 50 συν σε ό,τι αφορά την επισφάλεια στην αγορά εργασίας. θα πρέπει να ε, δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ε, εκπαίδευση ψηλής ποιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανώτερη εκπαίδευση, μια εκπαίδευση που θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ε, αγοράς εργασίας. Η σχετική τροπολογία για την κατάρτιση που θα πρέπει να έχετε σε σύζευξη με τη, ζήτηση της αγοράς εργασίας είναι κάτι που κινείται στη δική μου λογική. Πρέπει πραγματικά να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα άτομα που δυσκολεύονται ουσιαστικά να έχουν πρόσβαση στην αγορά και να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν τα κατάλληλα εφόδια. Η στήριξη λοιπόν που μπορεί να λάβουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές από το κοινωνικό ταμείο ε, είναι πολύ σχετική. και θέλω εν στο κείμενό σας να προσθέσουμε κάποιες αναφορές στην απλούστευση τη διαδικασία επιλογής των εταίρων στα σχετικά project ώστε να καταλήξουμε σε ένα πραγματικά πλουστευμένο σύστημα στο αφορά αυτή η διαδικασία. Είναι κάτι που απασχολεί όλους, πιστεύω, και τις μικρές οργανώσεις ε, και όλους μας, σε ό,τι αφορά τώρα τους διαγωνισμούς και τον τρόπο προκήρυξης διαγωνισμών είναι κάτι που μας απασχολεί χρόνια. Το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Δεν βλέπουμε όμως τελικά να γίνεται κάτι στην πράξη. Ένα άλλο θέμα που με απασχολεί είναι ε, το χάσμα στις απολαβές ε, ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Χρειάζεται μια σχετική τροπολογία, την οποία θα υποβάλω για να είναι πιο ξεκάθαρο το κείμενο προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά από πλευρά μου. Συγχαρητήρια πάντως στην εισηγήτρια για, την, ε, για το κείμενο αυτό. και πιστεύουμε ότι στην τελική του μορφή ο κανονισμός αυτός ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να στηρίξει περισσότερες και καλύτερες ποιότητας θέσεις εργασίας, κάτι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ύπαρξη και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια για τις τροπολογίες που έχει δηλαδή υπόψη και θα υποβάλω, όπως είπα, και άλλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Και τώρα κύριε Σρότερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που ξεκίνησε από πολύ νωρίς και διευκόλυνος εκ τούτου και την κατάθεση των τροπολογιών. Κάποια σημεία επί της ουσίας μας απασχολούν και θα θέλω να το αναφέρω γιατί στο θέμα των περιφερειακών αρμοδιοτήτων και μη περιφερειακών αρμοδιοτήτων, το τι είναι δηλαδή περιφερειακές αρμοδιότητες και τι μη. Εγώ Φερρυπίν θεωρώ στις ε, περιφερειακές αρμοδιότητες είναι το να ζητεί μια επιχείρηση ε, στην ευρύτερη περιφέρεια να ε, βρει εργαζομένους και να ζητήσει σε αυτό βοήθεια. Ίσως έχουμε διαφορετική εκτίμηση στο θέμα αυτό από τη γραμματεία για το κατά πόσον πρόκειται για περιφερειακό ζήτημα. Και ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι, σε κάθε, ότι η λέξη περιφερειακός δεν υπάρχει σε όλες τις τροπολογίες. Δηλαδή, εάν αλλάξει ένα σημείο του κανονισμού ο όρος αυτός και προσαρμοστεί, τότε θα πρέπει και οι λοιπές ε, ε, τα λοιπά εδάφια του κανονισμού που αναφέρουν την ίδια διατύπωση να προσαρμοστούν αναλόγως ε, για να μην υπάρξει παρεξήγηση, παρερμηνία. Γιατί διαφορετικά μπορούμε να έχουμε ε, μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία ξεκινούν σε μια περιφέρεια, προσλαμβάνει μια επιχείρηση εργαζομένους, στη συνέχεια όμω κλείνει, πηγαίνει σε άλλη περιφέρεια και απολύει βέβαια τους εργαζομένους. Επομένω θα πρέπει να κοιτάξουμε και σε σχέση με την αξιοπιστία, σε σχέση με την ε, σχέση εμπιστοσύνη, πώς μπορούμε να ε, επαληθεύσουμε τα ζητήματα αυτά. Αυτό είναι ένα που μα απασχολεί επίση. Και ένα άλλο είναι το θέμα της συγκέντρωσης είναι περισσότερο διαρθρωτικό ζήτημα. Η εισηγήτρια στις ε, τροπολογίες της έχει καλύψει ένα βαθμό και μετά τις συζητήσεις τις προτάσεις αυτές, τις ιδέες αυτές. Έχω κάνει και εγώ τις προτάσεις μου με τροπολογίες. Το θέμα είναι λοιπόν και θεματολογικά πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα της συγκέντρωσης. Σε επίπεδο προτεραιοτήτων για επενδύσεις. Και έχω ουσιαστικά στην τροπολογία μου ε, χρησιμοποιήσει την ορολογία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για το Κοινωνικό Ταμείο και επικεντρωνόμαστε όπως και στο ΕΤΠΕ σε τρία επίπεδα. Έχουμε δώσει έμφαση σε ένα θέμα που έχει και το earmarking βέβαια, δηλαδή την φτώχεια, την αντιμετώπιση της φτώχειας και προχωρούμε εκ παραλλήλου με την προσπάθεια αυτή. Ε, οι δείκτες και ο προσδιορισμός των δικτών είναι ένα δύσκολο θέμα, διότι η Επιτροπή είναι σε μεγάλο βαθμό προσεκτική ε, σε σχέση με τους δείκτες. Αφετέρου όμως ήταν και ασυνεπής. Ε, βλέπουμε ασυνέπεια Δηλαδή αναφέρεται σε ένα σημείο σε δείκτης, αλλά όχι παντού. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει, σε αυτό θα πρέπει να γίνει τροπολογία για να εξασφαλιστεί ε, συνέπεια. Ξέρουμε ότι έχουν διαφορετική στάση φερειπίνη στο θέμα των ανδρών και γυναικών ε, οι επιχειρήσει. Εγώ το έχω δουλέψει πολύ το θέμα αυτό, τα έχω καταγράψει και σε βιβλίο. Άρα λοιπόν θα ήθελα να δημοσιεύονται στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο μια γυναίκα επιχειρηματίας, μια γυναίκα που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, αντιμετωπίζει ε, ζητήματα οργανωτικά ε, και πώς δυσκολεύεται να επικοινωνήσει ακόμη και με υπουργούς και δύο, όχι άντρες, αλλά γυναίκες δυστυχώς. Άρα λοιπόν το θέμα της επαλήθευσης προς το φύλλο θα πρέπει να το ε, εισαγάγουμε σε κάθε σημείο του, του, του κανονισμού, όχι σε ορισμένε μόνο διατάξει. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κάτι άλλο που έχει σημασία για το άρθρο 5, γιατί είναι σημαντικό για το γενικό κανονισμό, εταιρική σχέση και ο τρόπος με τον οποίο δίνεται η χρηματοδότηση. νομίζω ότι έχει γίνει ένα λάθος εδώ. Το σημείο 6 στο κοινωνικό ταμείο δεν αφορά μόνο εταίρους, αλλά διαφορετικές μορφές υλοποίησης του κοινωνικού ταμείου. Και άρα χρειάζεται για τους συντρόφους μια διαφορετική χρηματοδότηση. Και ο θεματικός στόχος 11 πάλι θα πρέπει να προβληθεί πιστεύω. θα είχε νόημα να συμπεριληφθεί μέσα στο κείμενο. Και να προτείνονται παράλληλοι δρόμοι, διότι βέβαια δεν είναι πάντοτε ισότιμες οι μέθοδοι που εφαρμόζει η διοίκηση για να χρηματοδοτεί του, τις δραστηριότητες των κοινωνικών εταίρων Φερρυπίν. Άρα ναι, πρέπει να υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι. Δεν είναι απαραίτητο να αιτιολογείται καν το ότι υπάρχει ενδεχομένω διαφορετική στάση ή μέθοδος από πλευράς των κρατών μελών, γιατί κάθε κράτος μέλος μπορεί από τις δύο ή, αυτε, ή τρεις αυτές μεθόδους που προβλέπονται να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. Αυτό που λέμε εμείς όμως είναι ότι διατυπώνεται ένας κανονισμός για τους πάντες, έτσι. Και ανάλογα με τις εθνικές ιδιαιτερότητες αξιοποιείται και υλοποιείται. Αυτές θα είναι οι δικές μας τροπολογίες. Απλώς θα πρέπει να σκεφτούμε πόσο σκόπιμες είναι ορισμένες από τις τροπολογίες που θα θέλαμε να καταθέσουμε και να τις συζητήσουμε. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ την συγκεκριά για την πολύ καλή συνεργασία. Σας ευχαριστούμε και περιμένουμε με χαρά τις τροπολογίες σας κυρία Σρέντερ και κυρία Ernst. Εδώ, όχι. Δεν είναι εδώ. to the rapporteur again for final remarks. Θα δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια τις ε, καταληκτικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. Οι δύο σκιώδεις συνεισέφεραν σημαντικά για τη βελτίωση αυτού του μέσου που και εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως εν καιρό κρίσης οι υποδείξεις σας και η συνεργασία, η διαπεριφερειακή, η διεθνική. Θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να είναι μάλιστα υποχρεωτική, αν θέλουμε το τάμενο να είναι αποτελεσματικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τους ε, ανθρώπους πάνω των 50 ετών, που είναι ενεργό κεφάλαιο, πράγματι πρέπει να τους παράσχουμε ε, βοήθεια. Επίσης, ε, η εκπαίδευση, η κατάρτιση για την προσαρμογή στην αγορά εργασίας, απλούστευση διαδικασιών και αυτό είναι πολύ σημαντικό δεν θα πρέπει να χάσουμε ώρα με τις λεπτομέρειες. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες και τις ε, προτάσεις της κυρίας Σρέντερ, να πω ότι κάποιες από αυτές είναι σκέψεις ε, που αφορούν τη διαδικασία και νομίζω ότι υπερβαίνουν αυτό το οποίο εγώ θα επιθυμούσα και ε, υπέβαλε και κάποιες ερωτήσεις προς τη γραμματεία για τη διαδικασία, το πεδίο εφαρμογή, ε, κατά πόσον πρόκειται για περιφερειακή αρμοδιότητα ή όχι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση, θεματική συγκέντρωση, αυτά τα συζητήσαμε και για τις προτεραιότητες ε, στις επενδύσεις. Όταν εκπονούσα αυτήν την έκθεση, ο στόχος μου ήταν πιο πολύ να μην αλλοιωθεί η φύση του Ταμείου αυτού. Θέλουμε να το ενισχύσουμε το πολύ σημαντικό αυτό εργαλείο, να το βελτιώσουμε, να το επικαιροποιήσουμε με τους δείκτες για να γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση. Νομίζω ότι μέσω του Κοινωνικού Ταμείου μπορεί να βελτιωθεί και η αγορά εργασία. Θέλουμε επίσης και αυστηρή εφαρμογή της χρήση και διαφάνεια με τη συνεργασία όλων των συναδέλφων πιστεύω ότι θα συνεισφέρουμε στο ότι το πολύ σημαντικό ήδη αυτό ταμείο θα αποδεί ακόμη πιο χρήσιμο, όπως είπα, σε καιρό κρίσης, όπως αυτό που βιώνουμε σήμερα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρίγκο Γιάννη Πέρες για τις παρατηρήσεις σας. Κύριε Σούκοβα τώρα από την Επιτροπή εάν έχω προφέρει σωστά το όνομά σα με συγχωρείτε. Αλλά μια και έχουμε τόσο περιορισμένο χρόνο, αν μπορείτε να περιορίσετε σε δύο λεπτά μόνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φυσικά, αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε τις ε, προτάσεις ε, σε κάποια άλλη στιγμή, έτσι πιο αναλυτικά. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες υποδείξεις, τις ε, στηρίζουμε πιστεύουμε ότι θα στηρίξουν, θα ενισχύσουν την πρόταση που σας ευχαριστώ που την υποστηρίζετε στις γενικές της γραμμές. για τους δείκτες που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, ίσως θα μπορούσαμε να τους επανεξετάσουμε και θα δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα και αν μετρώνται καλά. Δεν θα επαναλάβω γιατί επιλέγουμε τη θεματική ε, συγκέντρωση στις επενδύσεις, προτεραιότητες επενδύσεων και όχι σε θεματικούς στόχους. Η κυρία Σρέντερ λέει να επικεντρωθούμε αποχρωτικά στην αρχή της συγκέντρωσης από ό,τι κατάλαβα Στηρίζουμε επίσης ε, το ότι θα πρέπει οι τοπικοί περιφερειακοί ε, φορείς, μη καπάμικρο, να συμμετέχουν πλήρως στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Κοινωνικού Ταμείου. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Διοντολογίας είναι ένα καλό εργαλείο για να μπορέσουμε να αποκριθούμε σε αυτή την επιθυμία. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και αργότερα σήμερα και αύριο μπορούμε να είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε αναλυτικότερα κάποιες από τις προτάσεις μας που ίσως να είναι λίγο πολύπλοκες. Καλό θα ήταν να τις αναθεωρήσουμε για να μπορούν να εφαρμόζονται απλουστευμένα, με απλουστευμένο τρόπο. Αυτό το έχουμε ήδη ε, ακούσει ε, και σε κάποιες από τις ομιλίες των βουλευτών. Είναι σίγουρα ένας κοινός στόχος. Ja, herzlichen Dank für die präzisen Anmerkungen. Ich möchte Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ συγκεκριμένε σας απαντήσεις. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 31η Μαΐου στις 8, στις 6 το βράδυ. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε να δούμε και άλλες πολλές προτάσεις για το κοινωνικό τομείο. Ασφαλώς και από τη δική μου την ομάδα. Θα υπάρξουν προτάσεις και τώρα περνάω στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Μακροπεριφερειακές στρατηγικές και Εισαγωγικά παρακαλώ τον κύριο Αλφόνση να λάβετε το λόγο. Παρακαλώ κύριε Αλφόνση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μακροπεριφερειακή στρατηγική ξεκίνησε στην ε, Βαλτική, επικυρώθηκε το 2009 και η Κομισιόν λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή τη ε, μορφή συνεργασία ε, που πλέον επεκτάθηκε και στην περιοχή του Δούναβη, στη λεκάνη του Δούναβη. Θεωρώντα ότι με αυτή τη μακροπεριφερειακή συνεργασία ανοίγονται νέοι δρόμοι για μια πολιτική συνοχή στην Ευρώπη. Θέλαμε λοιπόν να έχουμε αυτή την εδαφική, αν θέλετε, ανάπτυξη. Ξέρουμε ότι το διεθνικό σκέλο θέλει η Κομισιόν να ενισχυθεί για να στηριχθούν νέε μακροπεριφερειακές πολιτικές και υπάρχουν και διάφορες προτάσεις μακροπεριφερειών. Θα πρέπει να συντονίσει η Κομισιόν, να εξασφαλίσει τη βιώσιμη διακυβέρνηση, να ορίσει κοινού και μετρήσιμους δείκτες. Επίσης, προτείνει η έκθεση να εγκρίνουμε τη μακροπεριφερειακή προσέγγιση της πολιτικής εδαφικής συνεργασίας διότι εκτιμά ότι τα σχέδια δαυκής συνεργασίας θα έχουν μεγαλύτερη ε, ε, υπεραξία, θα έχουν προστιθέμενη υπεραξία. Αξία, συγγνώμη. Επίσης, από κοινού πιστεύουμε ότι θα εξασφαλίσουμε και μια συνέργεια με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική μεταξύ άλλων. Και θα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά μέσα όπως αυτά της Τράπεζας Επενδύσεων. Η μακροπεριφερειακή συνεργασία θα πρέπει να έχει και τη συμμετοχή του τοπικού περιφερειακού επίπεδου και να δίνει στις πολιτικές ε, γειτονίας, στις προτεξιακές πολιτικές ε, επίσης ε, χώρο γιατί μπορούμε να αποκομίσουμε ωφέλη. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο μας έχει ψηφίσει μια πίστοση οικονομικής βοήθειας για τη Βαλτική, κάτι άκρος χρήσιμο για να μπορέσει να πηχθεί αυτή η στρατηγική και νομίζω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και για την λεκάνη του Δουνάβεως, ώστε η στρατηγική αυτή να λάβει την ίδια στήριξη και να έχει την ίδια τακτική παρακολούθηση και να έχει και κατάλληλη χρηματοδότηση. Μελλοντικές τώρα ε, ε, στρατηγικές, μακροπεριφερειακές όταν έχουμε τέτοιες προτάσεις θα πρέπει να τις ε, βλέπουμε συνολικά. Είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει με έναν χάρτη μακροπεριφερειών. Δεν νομίζω ότι η στρατηγική χρειάζεται νέου πόρους, ούτε νέα θεσμικά μέσα, ούτε νέα ρύθμιση κανονισμού. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι βοήθεια ε, με πόρους, τεχνικής βοήθεια ουσιαστικά. Η έκθεση αυτή, μεταξύ άλλων, προβάλλει τη σημασία της περιοχής της Μεσογείου στην Ευρώπη από αρχαιοτά των χρόνων, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά πρέπει να επανερχόμαστε γιατί η μακροπεριφερειακή προσέγγιση σε αυτό το ζωτικό για το μέλλον της Ευρώπης χώρο θα μπορούσε να ορίσει ένα συνολικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε έξοδο από τη σημερινή κρίση. Και έτσι ε, θα ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες των γειτονικών χωρών, ιδίως από την Νότια Αφρική. Η Μεσόγειος είναι ένα σύνολο συνεκτικό. Ίδια είναι η περιβαλλοντική και πολιτιστική λεκάνη, ίδια τα χαρακτηριστικά, το μεσογειακό κλίμα, γεωρικές καλλιέργειες, ε, υδάτινη ε, πόρη, ανανεώσιμες πηγές, ιδίως ηλιακή ενέργεια, τουρισμός πολύ σημαντικός, κίνδυνοι φυσικών καταστροφών ε, παρόμοιοι κτλ. κτλ. Η Μεσόγειος λοιπόν, ε, μια ευρύτατη περιοχή, Έχουμε τώρα το σχέδιο μακροοικονομικής στρατηγικής, έχει προχωρήσει και εγγράφεται σε μια μακρά παράδοση συνεργασίας και αλληλεγγύης. Προτείνεται λοιπόν η Κομισιό να στηρίξει την ιδέα της υλοποίησης μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Μελεκάνη της Μεσογείου και αυτή η στρατηγική θα πρέπει να δώσει στο Ευρωπαϊκό Τμήμα της Λεκάνης της Μεσογείου ένα δομικό, ισχυρό δομικό πλαίσιο το οποίο θα καταστεί προσβάσιμο και στις προενταξιακές χώρες και στις γειτονικές χώρες από την αλλιόχθη της Μεσογείου ώστε να βελτιωθεί η επιχειρησιακή δαφική συνεργασία μεταξύ των δύο οχθών της Μεσογείου. Θα πρέπει να εγκριθεί η στρατηγική αυτή γρήγορα από το Συμβούλιο και θα πρέπει να υλοποιηθεί μια συνολική στρατηγική στη Μεσόγειο. Αυτή θα βασίζεται σε πρώτο και στη Δυτική και στην Ανατολική Μεσόγειο και όλες αυτές οι ε, πρωτοβουλίες θα πρέπει να συντονίζονται για να έχουμε μια συνολική εικόνα για τη λεκάνη της ε, Μεσογείου. Αυτή η συνολική εικόνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέργειες με τις προτεραιότητες που έχουν ορίσει οι διεθνείς περιφερειακές οργανώσεις και ιδίως η Ένωση για τη Μεσόγειο. Για να ολοκληρώσουμε, θεωρούμε ότι είναι καιρός ε, να αποφασίσει από αυτού το Κοινοβούλιο, ψηφίζοντας την έκθεση, ώστε να στηρίξουμε την ε, συνεργασία που βλέπουμε να αναδύεται στη λεκάνη της ε, Μεσογείου το επόμενο εξάμεινο, δηλαδή ε, η Κυπριακή Προεδρία ε, είναι θετικό γιατί η Κύπρος είναι στη Μεσόγειο ε, και ελπίζουμε ότι και η Κύπρος θα προωθήσει αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Ακούσαμε τον εισηγητή, σας από τους Σκιώδης. Παρακαλώ εσείς. Κύριος Δόιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον κύριο Αλφόνση για το σχέδιο εκθέσεως και να κάνω κάποια συγκεκριμένα σχόλια, αν επιτρέπετε, για την έκθεση αυτή. Καταρχάς, συμφωνώ ότι η μακροοικονομική στρατηγική, μακροπεριφερειακή στρατηγική, όπως και η στρατηγική για τον ε, Δούναβη, είναι πολύ σημαντικές διστάσεις της περιφερειακής πολιτικής και οι στρατηγικές ανοίγουν νέα κεφάλαια στην ε, ιστορία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ προσωπικώς συμφωνώ με τον κύριο Αλφονσί ότι χρειάζεται μια αξιολόγηση γερή, μια αξιολόγηση σθέναρη, όχι μόνο γραφειοκρατική και για τη στρατηγική της Βαλτικής. Και πρέπει να δούμε αποτελέσματα αυτής της στρατηγικής και να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες σε σχέση με τη στρατηγική για τη Βαλτική, να επικεντρωθούμε στους στόχους και τις ε, προσπάθειες που έχουν γίνει. Συν το χρόνο θα πρέπει να αξιολογήσουμε και την ε, λειτουργία της στρατηγικής για το στις ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές του μέλλοντος βλέπουμε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία, ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο που θα αναπτυχθούν αυτές. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι. Μερικές φορές αντιφατικές μεταξύ τους αποτελέσματα. Για δε τη στρατηγική, για τον ε, για την ε, Βαλτική, έχει μεγάλη σημασία αυτές οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές να εξασφαλίζουν συμμετοχή ευρεία φορέων με κυβερνητικών οργανώσεων, ενδιαφερομένων παραγόντων και πολυκυβερνητική μέθοδο και όχι διακυβερνητική. Έτσι καταλήγουμε σε πολύ συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και ως εκ τούτου είναι προφανές ότι εάν θεσπίσουμε κριτήρια, ένα σύστημα με κριτήρια ή αν ε, συγκρίνουμε με τις προηγούμενες πρακτικές Δηλαδή, αν όπως στο παρελθόν θεσπιστούν αυτέ τι στρατηγικέ μόνο για λόγου πολιτική επιλογής, τότε δεν θα έχουμε σωστά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι ο χάρτη των, υπερ, των ε, μακροπεριφερειακών στρατηγικών, αυτή η ιδέα τη Επιτροπής, είναι ενδιαφέρουσα. Εάν δεν υπάρχει χαρτογράφηση πάντω και δεν υπάρχει αξιολόγηση προηγουμένων στρατηγικών, θα είναι πολύ δύσκολο να διαγράψουμε και τις στρατηγικές στο μέλλον. Εγώ υπογραμμίζω βέβαια τη στρατηγική για τη Μεσόγειο. Δεν θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι μιλούμε για τρεις ή τέσσερις διαφορετικές μακροπεριφερειακές στρατηγικές αυτή τη στιγμή. Και καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει η εικόνα και με πολύ σαφή τρόπο να διαγραφεί μια κοινή θέση είναι απαραίτητο πιστεύω να διευκρινιστεί ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί. Εν τέλει δε, για την προσεχή δημοσιονομική περίοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μπορεί να γίνει επέκταση του προϋπολογισμού για την εδαφική συνεργασία από 2,5% δηλαδή, να αυξηθεί το ποσοστό στο 3,5% είναι πολύ σημαντικό πιστεύω να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν, να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλα οι πόροι που χρειάζονται. Και αυτό να το μεταφράσουμε και σε πράξη και στο μέλλον, γιατί συνεπάγεται, σημαίνει προσθέμενη αξία και βελτίωση στην εδαφική συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την έκθεση και βεβαίως θα υποβάλω και εγώ κάποιες τροπολογίες για να τις συμπληρώσω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καρόνα εδώ. Κύριος Δε Άντζελης θα αναλάβει νομίζω, αλλά παρακαλώ πάλι όλοι όσοι λαμβάνουν το λόγο να είναι σύντομοι. γιατί ακολουθούν και άλλες δύο ακόμη εκθέσεις. Παρακαλώ. Κύριος Δεάντζελης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας μεταφέρω την ε, συμβολή του συναδέλφου του κύριου Καρόνα που δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας εξαιτίας του σεισμού ε, που έπλεξε την Ιταλία και την περιφέρεια της Εμίλιας. Να πω τώρα στην ουσία. Ευχαριστούμε και εμείς τον ε, συνάδελφο για την έκθεση, η οποία έχει λάβει υπόψη ε, πολλά από τα θέματα που συζητήθηκαν το περισμένο διάστημα και σε ό,τι αφορά τις ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές, οι υπόθηκε, έχουν δώσει μια σημαντική ευρωπαϊκή προσιδέμενη αξία. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτή ακριβώς την πορεία ελπίζουμε το Συμβούλιο και η Κομισιόν να εξεύρουν αντίστοιχες ε, στρατηγικές και σε άλλους τομείς. Αυτές οι στρατηγικές θα πρέπει να κινηθούν όμως σε σαφώς προδιαγεγραμμένες γεωγραφικές περιοχές. Και μάλιστα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, για να θέλει το να είναι η λειτουργικότητα και η συνεργασία, η προσέγγιση θα πρέπει να είναι ότι έχουμε εδαφική διαφυριπηριακή συνεργασία για να δώσουμε και προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα του πολίτη. Πράγματα που χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Μεσόγειο, βλέπω θετικά αυτή την πρόταση για μια στρατηγική της δυτική Μεσογείου, όπως και για τις ε, Ανατολικές Λεκάνες. Δηλαδή αναφερόμαστε στο Ιόνιο Πέλαγος και την Ιδρυατική Θάλασσα α, τελευταίο διάστημα έχει καταδειχθεί πραγματικά ότι είναι ε, μία περιοχή σημαντική για την οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια στρατηγική μακροπεριφερειακού χαρακτήρα. Πολύ ορθά λέγεται ότι η Μεσόγειος έχει ιδιαίτερα χρηστικά και τα δικά της προβλήματα. Ο τρόπος όμως ε, με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, τα ιδιαίτερα προβλήματα των δύο ε, θαλάσσιων λεκανών ε, δεν μπορεί να γίνει ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των θαλάσσιων αυτών λεκανών. Έπειτα κάποιες τροπολογίες που ελπίζουμε να πλουτίζουν το κείμενο. Αναφερόμαστε στην περιοχή της Ατρετικής και του Ιωνίου Πελάγους και ελπίζουμε να δεχτούν αυτές τις τροπολογίες στο Συμβούλιο και Κομισιόν ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί μια μακρο ε, οικονομική στρατηγική για αυτή την περιοχή της Μεσογείου όπως έγινε αντίστοιχα με την ε, Δυτική Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ευχαριστώ και Δημοκρατών τώρα, ε, μάλλον ε, τώρα έχουμε τους φιλελευθέρους, αλλά δεν βλέπω την κάρτα σας καλά και δεν μπορώ να διαβάσω το όνομά σας. Αγκαίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος ε, Ούτσας, ως κοιόδης εισηγητής ε, για την ε, ομάδα των φιλελευθέρων, θέλω να εκφράσω τη στήριξή μου, την υποστήριξή μου, συγγνώμη, έναντι της έκθεσης Αλφονσή και ειδικά αυτή την πρόταση για μία μακροοικονομική στρατηγική για την Μεσόγειο, Ανατολική Μεσόγειο. Θεωρώ ότι έκανε μια εξαιρετική δουλειά ο εισηγητής. Μια δουλειά που χαρακτηρίζεται από πάθος και ιδιαίτερη προσοχή σε πολλά επιμέρους σημεία. Θέλω να ασχοληθώ σε αυτή μου την παρέμβαση για ένα ειδικό συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν θέλω δηλαδή να επαναλάβω τα γενικά ζητήματα, γενικά εκτεστικά, τα γενικά επιχειρήματα που ήδη εξέφρασαν οι προλαλήσαντες. Ξεκινώ από το εξή γεγονό, την εξή σκέψη, ότι η λεκάνη τη Μεσογείου είναι μια πολύ εκτεταμένη γεωγραφικά περιοχή και ποικίλει σε πολλά στοιχεία. Ο εισηγητή, μάλιστα, προσπαθεί να κάνει μια υποδιέρεση της Μεσογειακής Λακάνης σε τρεις ε, γεωγραφικές περιοχές. Ανατολική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος και Κεντρική Μεσόγειος, δηλαδή Εδρετική και Ιόνιο Πελαός. Όπως ε, ακούστηκε πριν από λίγο, αυτή ε, η γεωγραφική, τελευταία γεωγραφική περιοχή αυτή τη στιγμή ε, προσδιορίζει τα καλύτερα και είναι στη φάση τελικής, αν θέλετε, διαμόρφωσης. Πρέπει να κάνουμε, ε, πιστεύω, και μία προσθήκη ακόμη. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για μία για τον ισιωτικό χώρο της Μεσογείου. Δηλαδή μιλάμε για τη Μεσόγειο γενικά, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε και στα νησιά που θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς για μια ειδική πολιτική. Μια πολιτική που θα μπορούσε να αφορά τα νησιά της Μεσογείου, αλλά όχι και μόνο αυτά. Η Κομισιόν έως τώρα δεν ε, θεώρησε σκόπιμο να εξειδικεύσει πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές. Και αυτό βασίζεται γενικά και αόριστα στο ότι είναι πολύ μικρό ο πληθυσμό σε σχέση με το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να εστιάσουμε να εξειδικεύουμε σε αυτό το βαθμό. Ε, ε, ε, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε όμω επί τη ουσία αυτό το ζήτημα. Πώ δηλαδή οι νησιωτικέ περιοχέ αντιμετωπίζουν διαρθρωτικά handicap. Πλήγεται από τέτοια handicap, ελλείμματα διαρθρωτικά, Ακριβώ γιατί ζουν μια μορφή απομόνωση λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας μιας νήσου και άρα απαιτούν μια ειδική στήριξη από την πολιτική συνοχή. Αν δεν είμαστε εμείς εδώ, σε αυτό το βήμα που μιλούμε για την περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική και δεν θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη το πρόστο κόστος των πρώτων υλών, της ενέργειας, τη λιγότερη προσβασιμότητα στην ενιαία αγορά και τις νησιωτικές περιοχές, τότε πιστεύω ότι σφάλουμε. Σφάλουμε σημαντικά έναντι των των κατοίκων αυτών των ισιωτικών περιοχών. Θεωρώ λοιπόν ότι η προστίκη μιας τέτοιας ειδικής κατηγορίας και εδώ θέλω να προκαταλάβω και μια σειρά τροπολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τι μεταφορέ, τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας και μια σειρά άλλων θεμάτων, μπορούμε να εξειδικεύσουμε περαιτέρω μέσα από αυτή την έκθεση για τις μυστικέ περιοχές Και τέλος αλλά σημαντικό, είναι το εξή. Γενικά, σε αυτό το φάκελο, σε αυτή την έκθεση, θα πρέπει να μπει η λογική μιας, ενός στρατηγικού, αν θέλετε, σχεδίου, που να δίνει ιδιαίτερη σημασία στο εξής ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις μακροπεριφέρειες και να υπάρχει μια ειδική πολιτική μακρο, ε, διακυβέρνησης ακριβώς βάσει αυτών των ειδικών αναγκών τους. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε από το βλέπω εδώ άλλους σκιώδεις. Αν δεν αντιδρά κανείς, κλείνω τον κατάλογο. Δεν είσαι σκιώδης Λαμπέρτ, ούτε, έχεις, ούτε είναι σειρά τώρα καθένας με τη σειρά. Μα πάτε πολύ γρήγορα φαίνεται. Ναι, ναι, αλλά θέλω να σας παρακαλέσω όλους να περιοριστείτε στο ένα 15 λεπτό. Δεν έχουμε χρόνο, δεν θα προλάβουμε. Πολύ σύντομα λοιπόν. Κυρία Λουκασέφισκα ξεκινάει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι πολύ καλή δουλειά που έκανε. Θα ήθελα επίσης να πω ότι υποστηρίζω τη θέσπιση μακροπεριφερειακών στρατηγικών, καθώς από ό,τι βλέπω προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα και σημαντική ευρωπαϊκή προσταμινή αξία. Πολλά είναι και τα προβλήματα πέραν των νέων πρωτοβουλίων που μπορούν να αναπτυχθούν. Πολλά είναι τα προβλήματα που μπορούν να επιληθούν ε, διασυνοριακά, ε, περιφερειακά, ε, περιβαλλοντικά ζητήματα, ζητήματα εκπαίδευση, δημιουργία θέσεων κατάρτιση. Άρα λοιπόν όταν έχουμε αυτήν την ε, κίνηση από κάτω προς τα πάνω, όταν υπάρχει αυτή η βούληση από τη βάση για συνεργασία, θα πρέπει πάντοτε να προσφέρουμε εμείς το πλαίσιο, το πλαίσιο για την θέσπιση μακροπεριφερειών. Και... Χαίρομαι ιδιαίτερα για την πρόταση για τη χαρτογράφηση των μακροπεριφερειών. Ελπίζω δε αυτοί οι χάρτες να είναι δεσμευτικοί και όχι μη δεσμευτικοί όπως αναφέρατε στην έκθεση. Ελπίζουμε επίση να προσφέρουν νέους, νέες μακροπεριφέρειες αυτός, αυτή η έκθεση. Και για να αφαιρθώ στη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, τα Καρπάθια όρη, η μακροπεριφέρεια πρέπει να πω ότι έχει στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία. Και ελπίζω ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία για καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Θα καταθέσω βέβαια και τις δικές μου τροπολογίες, αλλά ελπίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ε, την ε, πολιτική συνοχή στον συγκεκριμένο αυτόν τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ταχύτατα ο κύριος Σφανής Ρούι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ε, τάσομαι πολύ θετικά σε σχέση με την εκθέση αυτή. Κάποιες παρατηρήσεις που έχω να κάνω τις έχει εκθέσει ήδη ο κύριος Τόμας Δόιτς. Δύο παρατηρήσεις για να επανέλθω στην χρονική στιγμή κατά την οποία προσδιορίσαμε τις ε, θέσεις μας. με τον κανονισμό που δίνει μια ευρύτατη βάση και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό γιατί αναφερθήκατε και στην τεχνική βοήθεια, σε πολιτικά προγράμματα, που έχουμε ήδη από την εξωτερική πολιτική, αλλά στην διαπεριφερειακή, μάλλον στην εδαφική καλύτερα συνεργασία, έχουμε πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Και θα θυμηθώ και τα τρία όχι που είχαμε υπογραμμίσει, τα οποία δεν τα βλέπω πια, ίσως κάπου χάθηκαν. Τα όχι τι ήτανε, ήταν ότι δεν δεχόμαστε επιπλέον κονδύλια, δεν υπάρχουν μάλλον επιπλέον κονδύλια για δομές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν Ας τα υπενθυμίσουμε αυτά. Ας μην καλλιεργούμε ανεδαφικές ελπίδες, φρούδες ελπίδες. Πολλά μπορούν να γίνουν. Αλλά με την αξιοποίηση των υφισταμένων μέσων. Ούτως ή άλλως αυξάνεται και ο προπολογισμό. Έχουμε την εθνική συνεργασία, έχουμε την περιφερειακή συνεργασία. Υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης. Υπάρχουν σημεία από τα οποία μπορεί κανείς να αντλήσει πόρους. Έτσι, να τελευταία όλα αυτά αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Στην ευρωπαϊκή, λοιπόν, μακροπεριφερειακή χαρτογράφηση είναι η εντύπωση ότι θα μπορούσαν και να συμπίπτουν οι περιφέρειες, να υπάρχει δηλαδή επικάλυψη. Αυτός ο προτινόμενος χάρτης, τι ακριβώς μοίρα θα έχει, θα είναι α, πρακτικός, θα είναι ρεαλιστική επικόνηση που θα προσφέρει ή θα οδηγεί σε εσφαλμένες εντυπώσεις. Νομίζω ότι πρέπει μια τέτοια, ένα τέτοιο χάρτη με την, με την πρόταση του κύριου Αλφόνση να την έχουμε και να είναι ουσιαστική η για τον ε, χώρο της Μεσογείου Φεροπίνα, αλλά περαιτέρω δεν βλέπω τι μπορεί να προσφέρει. Πρόεδρος, ναι, πέραστε πάλι στο ε, ουσία θα πρέπει να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι πρέπει να περιοριστούν οι ομιλίες, οι παρεμβάσει σε ένα λεπτό. Ιδάλω δεν προλαμβαίνουμε να ακούσουμε τι άλλε τις τις ε, εκθέσεις. Λοιπόν, κυρία Λαντζόνη, και θα σας διακόπτω, σας Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να περισσότερο το 1,5 λεπτό. Εκτιμώ ιδιαίτερα αυτή την έκθεση. Συμφωνώ και εγώ ότι το θέμα αυτό είναι πολύ επικαιρό σήμερα. Η νέα πρόταση λοιπόν που υποβάλλεται για μια νέα στρατηγική μακροπεριφερειακή για τη Μεσόγειο θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρόταση. Υπάρχει μια πολιτική ευαισθησία για αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Είναι ένα παλαιό σχέδιο, ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Καλό είναι κάποια στιγμή να γίνει. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές αποτελούν ένα πρότυπο της χρήσης εφιστάμενων ε, εργαλείων, οπότε εγώ προσυπογράφω τον κανόνα των τριών όχι, όμως σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πολιτική συνοχή θα πρέπει αυτό να έχει μια προτεραιότητα, δηλαδή μια παρόμοια οργάνωση και χρήση αυτών των εργαλείων, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να μας οδηγήσει μια κατά προτεραιότητα χρήση αυτών των εργαλείων σε τέτοιου είδους στρατηγικές. Αυτή θα πρέπει να είναι η κοινοτομία, κατά τη γνώμη μου. Ιδάλω απλά αναμασάμε ε, ό,τι έχουμε πει εδώ και χρόνια. Βέβαια σου λέω ότι ο εισηγητής έχει μια τάση να κινηθεί σε τρεις διαφορετικές στρατηγικές για τη Μεσόγειο, ξεκινώντας, έχοντας ως πρότυπο παράδειγμα την ε, στρατηγική μακροπεριφερειακή για την Ιδρυτική και το Ιούνιο Πέλαγος, εγώ θα λέγω ότι διαφωνώ με τη μέθοδο που ακολουθείτε. Το να πολλαπλασιάζουμε στρατηγικές και να κατακαιρματίζουμε τις γεωγραφικές περιοχές δεν είναι κάτι καλό. Εντάξει, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σταματήσουμε και να μπλοκάρουμε τη στρατηγική για την Εδρετική και το Ιόνιο Πέλαγος, αλλά αντίθετα γενικότερα θα πρέπει να μην κατακαιρματίσουμε τη Μεσόγειο. Ιστορικός πώς μας στους αιώνες Μεσόγειος είναι μια ενιαία γεωγραφική περιοχή και έτσι θα πρέπει να τη βλέπουμε. Εντάξει, το ένα λεπτό το ξεπεράσατε, αλλά ας προσέχουμε από εδώ και προς κυρία Πέρες. Σύντομα, να πω και εγώ ότι ευχαριστώ κύριο Αλφονσέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε. Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξή σε διαφορά μας προλαλήσατες κάποια σημεία σημαντικά που θα πρέπει να λυθούν πάνω σε αυτή την έκθεση. Τι μου λείπει. Μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στη σημασία της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαφόρων μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Δεύτερον, πιο πολύ να δώσετε έμφαση στην πολυεπίπεδη κυβέρνηση και τη σημασία μιας πιο στενής συνεργασία, όχι μόνο των τοπικών και περιφερειακών αρχών αλλά και των διαφερομένων μερών του ιδιωτικού τομέα και των οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών λαμβάνοντας υπόψη ε, και ε, τα ενδιαφερόμενα ε, σχετικά δίκτυα προσωπούν ε, τους πολίτες. Έπειτα να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε έναν βιώσιμο τουρισμό που δίνει πόρους σε αυτές τις γεωγραφικές οχές και να προστατευτεί η βιοπικιλότητα της Μεσογείου. Τέλος, να επισημάνουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία του αστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της στρατηγικής μακροπεριφερειακού χαρακτήρα και να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην βιομηχανική ανάπτυξη, ιδίως αναφέρομαι στις λιμενικές περιοχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σάρα τελευταία για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ υποστηρίζω την ε, έκθεση του κύριου Αλφονσί Θέλω να κάνω κάποια επιμέρου σχόλια όσο γίνεται πιο σύντομα. Πρώτα απ' όλα θέλω να αποσαφηνίσω ότι αυτή η μακροπαυθερία θα πρέπει να δίνει προστιθάμενη αξία στα ήδη στα πράγματα που ήδη έχουμε και θα πρέπει να εστιάζει σε τομεί που θα βοηθήσει περαιτέρω να βελτιωθούν στην γεωγραφική περιοχή, ιδίω ό,τι αφορά τη διαχείριση ε, της, ε, του θαλάσσιου περιβάλλοντος προστασία του περιβάλλοντος ε, και μια όθηση περαιτέρω σε ανανεώσιμες πηγές και μια πολιτική υπέρ της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Θέματα κεντρικά και κομβικά για τη Μεσόγειο. Μια τροπολογία θα υποβάλλω σχετικά με τη στήριξη ε, στις νησιωτικές περιοχές και τις δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι σχετικές ε, περιοχές διότι πραγματικά πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα εμπόδια και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά στην προσβασιμότητα, ειδικά και στι μεταφορέ. Και κάτι παραπάνω για τον τουρισμό. Έχουμε να κάνουμε μια περιφέρεια που είναι ο πρώτο τουριστικό προορισμό ανά τον κόσμο και είναι κάτι που πρέπει να το πούμε και να το επισημάνουμε. Από εκεί και πέρα, καλή επιτυχία στον κύριο Φωνσή για το κείμενό του. Ευχαριστώ. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Κύριε Νίλσον. Όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Λφονσί για την εκθεσή του και για τα σχόλια βεβαίως που ακούστηκαν από τους ε, αξιότιμους ευρωβουλευτές να απαντήσω ειδικά στο ερώτημα του κυρίου Νόη κατά πόσον θα μπορούσαμε να έχουμε έναν ευρωπαϊκό χάρτη με τις μακροπεριφέρειες. κοιτάξτε, α, η, η συνεργασία μέσα από τις μακροπεριφέρειες έχει θελοντικό χαρακτήρα ε, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή βούληση και δέσμευση των κρατών μελών και των τοπικών περιφερειακών αρχών που δεσμεύονται για την ανάπτυξη και την υποστήριξη αυτών των μακροφεριών. Πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσαν κάποιες προτάσεις που ακούστηκαν σήμερα στη συζήτησή σας. Ιδίως ε, στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια, ε, τη Μεσόγειο που είναι μια τόσο μεγάλη γεωγραφική λεκάνη και κατά πόσο είναι καλό είναι να χωρίσουμε τη Μεσόγειο σε επιμέρους ε, περιφέρειες για καλύτερα αποτελέσματα. Το, το θέμα είναι πώς αυτές οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ε, και άλλες στρατηγικές που αφορούν τη διαχείριση ε, των θαλάσσιων πόρων και την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι πράγματι πρωτοβουλίες που ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποια πράγματα που λίγουν το 2014, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την απραγματικότητα. Ευχαριστώ. Okay, dann können wir das jetzt abrunden. Καλώς, μπορούμε να το κλείσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Αλφόντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους ε, όσοι εξέφρασαν την υποστήριξή τους και έδωσαν τη συμβολή του στην εκθέση. Αυτή δεν θα ε, υπησέλθω στην κάθε λεπτομέρεια των παρεμβάσεων. Είδαμε ότι εκδηλώνονται σαφές ενδιαφέρον για τη μακρό και στρατηγική από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί πρόκειται για μια στρατηγική η οποία είναι στη θέση να προβάλλει περισσότερο, αλλά και να δώσει περισσότερη ουσία στις πολιτικέ ε, πολιτικές ενταφικής ε, συνεργασίας. Για τον κύριο Φανίστηλ Ρόι θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι δεν απαιτούνται νέα δημοσιονομικά ή θεσμικά μέσα, ούτε και νέα ε, νομοθεσία, αλλά στηρίζεται σε επιστέωσεις τεχνικής συνεργασίας αυτή η μακροπεριφερειακή ε, στρατηγική. Άρα λοιπόν, για να μην αναφερθούμε με αυτήν την κάπως ε, λακωνική διατύπωση στα τρία όχι, τα αναφέρουμε ρητά. Και έτσι, όταν ορίζουμε ένα πλαίσιο πρέπει και να έχουμε υπόψη ότι κάθε μικροπεριφερειακή στρατηγική δεν έχει ε, τον ίδιο τρόπο υλοποίηση, δεν πρόκειται για την Βαλτική, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια ε, δυνατότητα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντονιστική, δυνατότητα να καταστήσει πιο ορατά τα προτινόμενα και για τους ενδιαφερομένους τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να προχωρήσουν από κοινού. Συνοχή δηλαδή στην εδαφική συνεργασία που υπογραμμίζεται, που εντοπίζεται ιδιαίτερα σε ζώνες με γεωγραφική κοινότητα, αλλά όχι πολύ συνοχή. Αυτά είχα να προσθέσω, ευπρόσδεκτες οι τροπολογίες. Το ζήτημα των νησιών φυσικά δεν έχω καμιά αμφιβολία και εγώ, άλλωστε το έθιξα ο ίδιος στην προηγούμενη έκθεση. Πρόκειται για ένα τα χαρακτηριστικά του χώρου της Μεσογείου και πιστεύω ότι με την υλοποίηση της έκθεσης αυτής και τη δουλειά που τη συνοδεύει, γιατί θα ήθελα να χαιρετήσω και όλες τις περιφέρειες, την Ένωση για τη Μεσόγειο, όλους όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την προσέγγιση αυτή. Ε, προχωρούμε λοιπόν σε ένα συνενετικό πλέον με έργο και σε μια δύσκολη χρονική στιγμή προσπαθούμε να ε, αντλήσουμε όλα τα θετικά μέσα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Λίγο ο Πρόεδρο. Και τώρα περνώ στο επόμενο θέμα τη ημερήσια διάταξη. Μάλλον πρέπει να πω προκαταβολικά ότι έχουμε ω προθεσμία την 1η Ιουνίου για την κατάσταση των τροπολογιών και έτσι περνώ στο επόμενο θέμα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής γνωμοδότηση amendments? Mm-hmm. Yes? Um, Sorry. No problem. Und hier haben wir als Berichterstatter für diese Opinion... Με ναι, εισηγητή, τον κύριο Ομάριε. Ελπίζω να προφέρω σωστά και το δικό σας όνομα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση, για τη σημαντική μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, η δική μας Επιτροπή έχει αναλάβει να εκπονήσει γνωμοδότηση. Ε, προσέχω λοιπόν τα μέτρα που προτείνω στην Επιτροπή μας ε, να είναι συμβατά βέβαια με την περιφερειακή πολιτική. Θέλησε επίσης τα, οι άκρως απομακρυσμένες περιοχές, περιφέρειες να μην ε, βρεθούν χαμένες, να μην ε, χάσουν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Ξέρετε ότι έχουμε χάρη σε αυτές τις άκρες απομακρυσμένες περιοχές τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη του κόσμου και άρα σε μια τέτοια πολιτική θα πρέπει και αυτές να μην λησμονηθούν, να μην μπουν στο περιθώριο. Καταρχάς και εν γέννη η νέα μεταρρύθμιση της κρίσης αλληλευτικής πολιτικής θα πρέπει να εγγυάται διαχείριση εγκύτητας, αποτελεσματικότητα στόλων, αλληλευτικών εξοπλισμών, θεμάτων προστασία σε κάθε χώρα και αλληλευτική ζώνη και εν γέννη αυτό είναι το των τροπολογιών που έχω καταθέσει. Επίσης απαραίτητο είναι να εξασφαλιστεί στις ε, παράκτιες περιοχές ε, στην Ευρώπη η βιώσιμη δραστηριότητα αλίας και υδατοκαλλιέργειας και γι' αυτό θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα στην υπεραλίευση για την περίοδο 2013-2020 και προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν για την απαιτούμενη ανασύσταση αλληλευτικών αποθεμάτων στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, μια τεράστια πρόκληση που ε, επιδιώκω να αντιμετωπίσω με μια σειρά από τροπολογίες όπως θα δείτε και αναφέρομαι βέβαια και στις επιπτώσεις για τον Αλία αλλά και για την επιμέρουσα περιφέρεια λέγοντας ότι αν δεν ε, πραγματοποιηθεί αυτή η προσπάθεια τώρα το μέλλον του ίδιου της Αλίας και η βιωσιμότητα οικονομική του κλάδου θα κινδυνεύσουν σοβαρά. Λυσμόνισα κατά την εισαγωγή μου να σας ε, παρουσιάσω το εξής αριθμητικό στοιχείο, ότι ο κλάδος της αλίας και της μεταπίεσης ελευμάτων αντιστοιχεί σε 350.000 ε, θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο σημαίνει σημαντική, σημαντικό ειδικό βάρος ε, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Πάντως, για την ανασύσταση των ολευτικών αποθεμάτων σημειώνουμε ότι αυτό θα πρέπει να προχωρήσει με τρόπο συνετό, γιατί κάθε ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική ε, δραστηριότητα που θα απορρεύσει από αυτήν θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά και βεβαίως με στόχο μακροπρόθεσμα να εξασφαλιστούν αξιοπρεπή εισοδήματα για τον αλιέα. Η οικονομική δυσπραγία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, οφείλεται θα έλεγα, σε εσφαλμένες επιλογές και των δημόσιων κρατικών αρχών. Και εδώ ε, πρέπει η κοινωνία να αναλάβει τις ευθύνες της. Δηλαδή δεν μπορεί ο αλλιέας να είναι ο μόνος ο οποίος θα πληρώσει το βαρύ τίμημα των εξελίξεων. Γι' αυτό λοιπόν η προσπάθεια δεν θα πρέπει να ε, γίνεται εις βάρος των αλλιέων και των οικογενειών τους, αλλά ούτε και εις βάρος των περιφερειών ε, που, είναι πιστρο, που έχουν τις αλληλευτικές δραστηριότητες ή εις βάρος των ε, συναφών δραστηριοτήτων. Αυτό το υπογραμμίζω και είναι απαραίτητο πιστεύω να εισαχθούν κανονισμοί, μηχανισμοί επιδότησης προσαρμογής για τους εργαζομένους στον χώρο της αλληλείας, που θα αντιμετωπίσουν τα σοβαρότερα προβλήματα σε οικονομικό, και κοινωνικό επίπεδο με σχέδια για ανασύσταση της πολιετούς διαχείρισης και καλύτερης ε, αντιμετώπισης και προστασίας των οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές για την αποκατάσταση των αποθεμάτων, για την αναθήσταση των αποθεμάτων και την βιώσιμη διαχείριση αποθεμάτων, ε, πόρων εισάγω και μία τροπολογία που υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στη διάσκεψη στην Αγκόια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεσμεύσεις για την θαλάσσια βιοπικιλότητα που λησμονείται συχνά. Εάν συνεχιστεί η υπεραλίευση με τους τωρινούς της ρυθμούς, μετά το 2050 δεν θα έχουμε ούτε ψάρι, ούτε μαλάκιο, στην ε, θάλασσα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει η εμπορική αλία. Μπορούμε να το ρισμόνουμε λοιπόν αυτό. Επίσης, ρητά τάσσομαι στην γνωμοδότησή μου κατά κάποιων προσπαθειών για εξασφάλιση δικαιωμάτων κυριότητας πάνω σε αλληλευτικά αποθέματα, δηλαδή εκχώρηση ε, μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων αλίας. Θα ήταν αυτό καταστροφή για την αλία και για τη διαχείριση των λευτικών αποθεμάτων, γενικότερα δε για τις περιφερειακές και, και θαλάσσιες ε, περιοχές μας και αυτό είμαι βέβαιος ότι βρίσκει συμφωνούς όλους τους αλείς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό πρέπει στο πλαίσιο της εμείς στην Επιτροπή μας να αντιταχθούμε στην πρόταση αυτή, πράγμα το οποίο προτείνω και με τις ε, τροπολογίες μου. Και τελευταία παρατήρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές και το υπογραμμίζω γιατί είναι και της Επιτροπής μας. Απαιτείται το άρθρο 341, απαραίτητο το άρθρο 341 για τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματωθεί στην μεταρρύθμιση αυτή και ρητά να αναφερθεί στον κανονισμό όπως κάθε μέτρο που εισάγει ε, παρεκκλήσεις. Ειδικότερα, θαλάσσιες λεκάνες όπου εργάζονται αλλοί των άκρων στους απομακρυσμένων περιφερειών που έχουν πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αντίστοιχες θαλάσσιες λεκάνες δεν αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο, γιατί τα, η κοινή αλευτική πολιτική στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στα χαρακτηριστικά της αλίας στο βόρειο ημισφαίριο. Επίσης, πρέπει να θεσπιστεί μία σειρά μέτρων ειδικών για τις άκρες απομακρυσμένες περιοχές. Αυτά λοιπόν σε μία πρόταση τα καλύπτω ζητώντας να ε, θεσπιστούν ε, συμβουλευτικές επιτροπές για τη διαμόρφωση νέων στόχων. Ιδιαίτερα για τις, υπερ... για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, αυτές θα δείτε ότι δεν συγκρίνονται ούτε με τη Μεσόγειο ούτε με την Βαλτική. Αυτό νομίζω δείχνει τις ιτερότητες αυτής της κατάστασης. Και θα ήθελα κλείνοντα πολύ σύντομα να πω ότι όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, οι τροπολογίες των συναδέλφων ε, και ότι η προθεσμία είναι πολύ σύντομη γιατί νομίζω μέχρι αύριο ή μεθαύριο έχουμε περιθώριο για κατάσταση τροπολογιών. Είναι ευπρόσδεκτες και παρακαλώ τον Πρόεδρο να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση των τροπολογιών για την γνωμοδότηση μου αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. όπω και στην προηγούμενη έκθεση, η 1η Ιουνίου προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Έχουμε ακόμα δύο μέρε, δηλαδή, δεν είναι όμω και πολύ ο χρόνο. Και Αποκλειστικά σε σκιώδει ηγητέ θα δώσω το λόγο. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Όχι, κλείνω και τον κατάλογο των ομιλητών. Και παρακαλώ και του σκιώδει να είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σύντομοι. Διαφορετικά θα προλάβουμε να συζητήσουμε το επόμενο θέμα. Και βέβαια το λέω αυτό και με σεβασμό στην δουλειά των διερμηνέων. Παρακαλώ λοιπόν. Ε, Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή σε ορισμένε από τι ανησυχίε που εξέφρασε με τι τροπολογίε του, ιδίω ό,τι αφορά τη πολιτική των απορρίψεων για τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Πιστεύουμε ότι το 2016 ε, θα είναι αβίωτη κατάσταση με την απόρριψη των ε, αλλιευμάτων. Θα πρέπει προοδευτικά να καταργηθεί αυτή η πρακτική. Βέβαια θα πρέπει ο στόλος να έχει και τον χρόνο στην ε, διάθεσή του για να μπορέσει να αλλάξει τα λευτικά εργαλεία που χρησιμοποιεί. Η βιώσιμη απόδοση είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, μια νέα παράμετρος που θα μπορούσε βέβαια να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στον αλληλευτικό στόλο. Η πρόταση πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνει επαρκώς υπόψη και τα συμπεράσματα του Johannesburg το 2012 στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εκεί έγινε λόγος για την ανάγκη να εφαρμοστεί αυτή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά μόνο στο μέτρο του δυνατού. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την εφαρμογή, ιδίως ε, σε κάποιες συγκεκριμένες ε, σε κάποια ακραία συγκεκριμένα αλλιεύματα. Για τη μεταβεβασιμότητα των αλληλευτικών δικαιωμάτων. Ο εισηγητή λέει ότι είναι αντίθετο με τη μεταβίβαση αυτών των αλληλευτικών δικαιωμάτων όπω προτείνει η Κομισιόν. Εμείς όμως υποστηρίζουμε στην προκειμένη περίπτωση την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντοτε βέβαια δίνοντα έμφαση στην ανάγκη να αποκλειστεί η παράκτεια μικρή κλίμακα ασαλία για να μην υπάρχει συγκέντρωση στους μεγάλους αλληλευτικούς ε, στόλους. Σε ό,τι αφορά τώρα τα πολυετή ε, προγράμματα, ο εισηγητής ε, λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένας κοινωνικο-οικονομικός στόχος για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις που θα έχουν στους θυγόμενους τομείς. Σε αυτό μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνο η άποψή του. Τώρα, για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε κάποιες από τις ε, φράσεις οποίες περιλαμβάνει η αλλά θα κάνουμε σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Μένα, δεύτερη συγγετρία, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Πάρα πολύ ε, η δουλειά του. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική βιώσιμη αλληλεία είναι σημαντικό πλεονέκτημα τη περιφέρεια. Έχουμε δει και γνωρίζουμε στην σημερινή αληφτική πολιτική ότι δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι τη βιωσιμότητα. Ε, άρα, εδώ πρέπει να πετύχουμε την αλλαγή. στους περισσότερους ε, ε, ψαρότοπου βλέπουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση να επικρατεί. Παραδείγματο χάρη στη Βαλτική, όταν οπολεύεται ο Σολομός, υπάρχει μεγάλο κίνδυνο, Αλλά είναι σημαντική αλία αυτή για τη Βόρεια Ευρώπη, για αεροκατοικημένες περιοχές. Δεν πρέπει να υπάρχει υπεραλίευση λοιπόν του Σολομού στο μέλλον, γιατί αυτό ε, θα είχε αρνητικές επιπτώσεις. Θα πρέπει ίσως να παγωρευτεί λοιπόν. Εγώ Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι καλό θα ήταν να πετύχουμε ε, την αποκατάσταση αυτών των ε, ψαροτόπων σε ένα βέλτιστο δυνατό επίπεδο και αυτό στο δυνατόν πιο γρήγορα. Ε, θεωρώ ότι ο στόχος αυτός έχει μια προθεσμία τεθεί το 2015 συγκεκριμένα. Είναι νομίζω κατάλληλη η προθεσμία. Ο σύγκριση προτείνει το 2017 δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι το 2015 είναι καλύτερα γιατί είναι πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα τι απορρίψει, η πρόταση να πάψει αυτό το φαινόμενο ε, τη Κομισιόν, η πρόταση μα βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Ευχαριστώ για την Επιτροπή, ίσως. Κύριε Νίκολσον, δεν είσαι στον κατάλογο, δεν σας έχω προβλέψει. Ναι, με είχα σηκώσει την κάρτα μου, αλλά ταυτόχρονα με τον άλλον ομιλητή και είμαι και σκιώδης ηγήτης εκ της ομάδας μου. I'm sorry, but you not on the list as shadow for, for this report. Δεν σας βλέπω στον κατάλογο των σκιώδων για την έκθεση αυτή. And... Yes, we don't have this group. It's not indicated this group. Okay. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί και η ομάδα μου μου είπε ότι θα είμαι σκιώδης για αυτήν την έκθεση και γι' αυτό είμαι εδώ. Okay, dann Καλά, τότε ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ τον εισηγητή για τις θέσεις του και τα σχόλιά του, τα οποία με βρίσκουν σε μεγάλο βαθμό σύντομο, γιατί είναι πολύ σημαντική ε, η μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα για τις απομακρυσμένες περιφέρειες και τις κοινότητες τους, ε, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ε, Συμφωνώ λοιπόν και υποστηρίζω την περιφερειοποίηση. Πρέπει να επανέλθει η περισσότερη εξουσία και αρμόδιότητες περιφέρειες στον κόσμο που δουλεύει εκεί και που ξέρουν ε, τι χρειάζεται. Επίσης πιστεύω ότι έχει σημασία να έχουμε μια πολυετή συμφωνία για το κόντι, για να έχουμε για τις ποσοστώσεις για να ξέρουμε τι γίνεται, δεν μπορεί κάθε Δεκέμβριο περιμένουμε να ληφθεί απόφαση για το τι είδους ποσοστώσεις θα ισχύσουν τον επόμενο χρόνο. Πρέπει αυτό να ανοησία που γίνεται μέχρι τώρα. Θέλουμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τις ποσοστώσεις. Θέσεις εργασίας, ε, χερσαίες ή θαλάσσιες και ε, απορριπτόμενα αλλιεύματα. Είμαστε εντάξει. Θα ήθελα να πω όμως για την μεταβίβαση των ποσοστώσεων ότι δεν θα πρέπει αυτές να επανέλθονται στα κράτη-μέλη. Πρέπει να πηγαίνουν στις πιο φτωχές και μικρές περιφέρειες. Και ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η άλλη κυρία των Πρασίνων παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προοπτική ε, υπό την οποία κινείται ο εισηγητής ε, και με τις που έχει και ο ίδιος σε περιλάβει είναι η εδαφική, ε, αν θέλετε, προοπτική. Έχετε δίκιο σε αυτή την προσέγγιση, γιατί δεν έχει ληφθεί διόντως υπόψη. Επίση, μιλάτε για την περιφερειοποίηση που συμμεριζόμαστε και εμείς ως ομάδα, αλλά αυτό που λείπει πιστεύω και αποδυναμώνει την έκθεσή σα είναι η ερασιτεχνική αλεία που αποτελεί και το 80% της δημιουργικής των Δηλαδή για να λάβουμε σωστά υπόψη ε, την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική συνιστόσα της αλείας, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις την ερασιτεχνική αλληλεία για τις ε, μελλοντικέ δεσμεύσει ε, θα υποβάλει σχετικέ ε, τροπολογίες, έλλειψη στατιστικών δεδομένων για τα επιστημονικά και κοινωνικά στοιχεία. Θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και οι τροπολογίες μπορεί να κάνει η Επιτροπή μας σε σχέση με τα επιστημονικά στοιχεία, τις απορρίψεις και την μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι ακριβώς ε, στοιχεία που κατά κύριο λόγο ε, απασχολούν την Επιτροπή Αλίας. Εμείς πιο πολύ θα πρέπει να μιλήσουμε για την βιωσιμότητα και την περιφερειακή βιωσιμότητα και, το πώς πρέπει να στηρίξουμε τις αλληλευτικές κοινότητες. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας συγγνώμη που είμαι έτσι πιεστικός τώρα και στο χρόνο. Δυστυχώς όμως δεν είχαμε άλλα περιθώρια και δεν μπορώ να δώσω και το χρόνο στον εισηγητή, στο συντάκτη για να απαντήσει. Είμαι βέβαιο ότι έχει κάνει, πάρει τι σημειώσει του. Για να προχωρήσω πάρα πολύ γρήγορα στα καινοτόμα χρηματοπροστατικά μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολίτη δημοσιονομικού πλαισίου, που είναι η επόμενη και τελευταία μα έκθεση. Η κυρία Κλέβα, η συγγετρία είναι παρούσα. Την παρακαλώ να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, ώστε να μην καταχραστούμε και του χρόνου των διερμηνέων. Θα είμαι σύντομη. Χρηματοδοτικά εργαλεία βάσει το νέο σύστημα είναι εργαλεία που στηρίζει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός που ε, επιτρέπουν να δοθεί μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο κινδύνου στις τοπικές οικονομίες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα εργαλεία ε, και γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε λίγα λεπτά παραπάνω στη συζήτηση για αυτή την έκθεση, γιατί ο στόχο είναι η επίτευξη των στόχων τη πολιτική συνοχή, η καλύτερη και πιο χρηστή, αν θέλετε, χρήση των κονδυλίων με την ενίσχυση της συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και συμμετοχή ενδιαφερμένων μερών. Οι επιδοτήσεις, οι χρηματοδοτήσεις, οι μικρο μικροχρηματοδότηση και όλα τα άλλα σχετικά μέσα που να χρησιμοποιηθούν. Βεβαίως ε, είναι πάντοτε έχουμε το ίδιο πρόβλημα, ότι δεν μπορούμε σε μία ε, γνωμοδότηση να βάλουμε τα πάντα, άρα θα πρέπει να κάνουμε μια γνωμοδοτηση να βαλουμε τα παντα αρα Θέλω να πω ότι στην περούσα κατάσταση, ε, σε μια εποχή δυσμενούς οικονομικής, αν θέλετε, συγκυρίας και σε εποχή λιτότητας, η χρήση αυτών των εργαλείων θα πρέπει να γίνει με τον πλέον καλύτερο τρόπο. Άρα να έχουμε επιχορηγήσεις, εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης και να να εγγυηθούμε κονδύλια για στρατηγικές επενδύσεις. Επίσης, ε, προσθέτω κάποια στοιχεία για την απλούστευση και την ε, σαφήνεια, πράγματα που τα γνωρίζουμε όλοι. Πρέπει να καταστήσουμε σαφή και στα θεσμικά όργανα και στις χειριστικές αρχές πριν την άνοιξη της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Θα πρέπει λοιπόν τα χρηματοδοτικά εργαλεία να είναι δελεαστικά, όχι μόνο για το δημόσιο τομέα, αλλά και τους ιδιώτες επενδυτές. Θα πρέπει να υπάρχει τεχνική ικανότητα για την χρήση και την διαχείριση αυτών των εργαλείων. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν ε, οι δημόσιες αρχές, οι ενδιάμεση και ιδίω οι τράπεζες. Έπειτα, η εκ των προτέρων αξιολόγηση. Κάτι που έρχεται και επανέρχεται στην Επιτροπή μα. Σε ό,τι αφορά αυτήν την αξιολόγηση, οι διαχειριστικέ αρχέ θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη χρηματοδοτικά εργαλεία εντοπίζοντα τα ελλείμματα και τι αποτυχίε στην αγορά και τι επενδύσει που δεν είχαν αποδώσει τα βέλτιστα αποτελέσματα και τέλο, σε ό,τι αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επόμενη πραγματική περίοδο και την πολιτική συνοχή θα, ε, θα πρέπει να διαχειριστούν σε όλους τους ε, θεματικούς στόχους. Κάτι που το οποίο χαιρετίζουμε. Όμως είμαι της γνώμης ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε μια σαφή εποπτεία της εφαρμογής αυτών των εργαλείων, ώστε να μπλύνουμε στο μέτρο του δυνατού ε, την έλλειψη τονισμού. Επειδή μας περιορίζει ο χρόνος, σταματώ εδώ και προσβλέπω στην εργασία με τους Κιώδη ε, για να κάνουμε τις καλύτερε δυνατέ τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση και τη στομία. Και τώρα έχω μόνο τον κύριο Φωνή στην Παρακαλώ, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, Πρέπει εδώ πραγματικά να αναφέρουμε και τα υφιστάμενα εργαλεία. Το Τζέσικα, τον τα λοιπά Πρέπει να εστιάσουμε στα κείμενα εργαλεία. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα πρέπει και οι εθνικές τράπεζες, οι ε, τράπεζες κρατών μελών να προσυπογράψουν αυτά τα νέα εργαλεία. Και βεβαίως θα πρέπει να μιλήσουμε ε, στο δυναμικό που απαιτείται από τους θεσμικούς φορείς των κρατών μελών. Μόνο έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, τη νέα δημοσιονομική περίοδο. Βέβαια είναι κάτι θα μας απασχολεί και θα εξετάζουμε κάθε χρόνο. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αποτελεσματικότητα βεβαίως, στη χρήση των κονδυλίων είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίω θα υποβάλουμε και τροπολογίε. Πάντω η έκθεση φαίνεται πάρα πολύ καλή. έχει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε και το θέμα αυτό. Άρα, σα ευχαριστώ πολύ όλου θερμά. Ευχαριστούμε του διερμηνεί και οι διερμηνεί σα ευχαριστούν. Χρειάστηκε να ξεπεράσουμε λίγο το χρόνο. Σα λέω ο πρόεδρο, αλλά τα καταφέραμε. Και Δεν έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα, εκτός από την ανακοίνωση ότι η προσεχής συνεδρίαση προβλέπεται για την 20η Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη και 21η Ιουνίου για τη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ, χαίρετε.